για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Η άδεια μητρότητας, αλλά και η γονεϊκή άδεια γενικότερα, η προστασία των εγγύων εργαζομένων και τα σχετικά θέματα είναι βασικά ζητήματα στην κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θεμελιωδώς σημαντικά για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής και κατά αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για μια αγορά εργασίας που θα λειτουργεί καλύτερα και για την καλύτερη χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, ο γενικός στόχος της Προεδρίας μας είναι το πώς θα μπορέσουμε να φροντίσουμε να δημιουργηθούν αγορές εργασίας πιο ανοιχτές προς όλους. Κατά τη γνώμη μας, οι δυνατότητες συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελούν ζωτική συνιστόσα προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να φροντίσουμε και οι μητέρες και οι πατέρες να μπορούν να συνδυάσουν την ιδιότητά τους ως γονείς και την ευθύνη τους για τα παιδιά τους με μια ισχυρή θέση στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η θετική επίπτωση της υψηλότερης συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην ανάπτυξη και την ευημερία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερος. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, των οποίων το ποσοστό απασχόλησης αυτή τη στιγμή είναι 14 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη πρόσβαση σε συστήματα που μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως ε, η φύλαξη των παιδιών ε, σε λογικές τιμές και συστήματα που λειτουργούν σωστά για την ε, ετήσια άδεια που έχει σχέση με την οικογενειακά θέματα, όπως επίσης και φορολογικά ζητήματα που ευνοούν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, είναι θέματα που μπορεί να βελτιώσουν τα ποσοστά απασχόληση των γυναικών και ακριβώ αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε. Η ισότητα των φύλων αποτελεί επίση προτεραιότητα τη Προεδρία μα και αυτό έχει σχέση με το θέμα των αγορών εργασία που είναι ανοιχτέ προ όλου, όπω είπαμε. Από αυτή την πλευρά πιστεύουμε ότι η οδηγία για την άδεια μητρότητας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και να συνεισφέρει στις ίσε ευκαιρίες για του άνδρες και τι γυναίκε στην αγορά εργασία. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τροπολογίες της οδηγίας αυτής περιλαμβάνει πολλές προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις εγγύους εργαζομένους και γυναίκες εργαζόμενες που ε, πρόσφατα έχουν ε, γεννήσει παιδιά. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι μεταξύ των κρατών μελών γενικά υπάρχει μια θετική άποψη όσον αφορά τι φιλοδοξίε μα να δώσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεσματικό για αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Βεβαίω από τι συζητήσει είναι σαφέ ότι διαφέρουν ε, αρκετά οι απόψει σχετικά με του τρόπου και τα μέσα για να το επιτύχουμε αυτό. Κάποια κράτη-μέλη λέγουν ότι η τρέχουσα οδηγία είναι επαρκής. Άλλα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για τροποποίησης, αλλά διαφωνούν όσον αφορά τους τρόπους και έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και συστήματα στα κράτη-μέλη σχετικά με τις διάφορες μορφές οικογενειακής άδειας και σχετικά με τα μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Αυτές οι παραδόσεις στα κράτη-μέλη είναι βαθιά ριζωμένες και στην κοινωνία και σε προσωπικό επίπεδο υπάρχουν διαφορετικές ατομικές απόψεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτέ τις διαφορές και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα με μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μπορούν να διατηρήσουν και να αναπτύξουν εθνικά συστήματα προστασίας των εργαζομένων, διαφορετικές μορφές οικογενειακής άδειας και την ισότητα των φύλων. Κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας, το Συμβούλιο καθόρισε ορισμένα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να βρούμε κοινέ θέσεις όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, άδεια μητρότητας. Είναι σαφές βεβαίως ότι χρειαζόμαστε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μας δώσει μεγαλύτερη όθηση και θα προωθήσει τις συζητήσεις μας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η Προεδρία περιμένει τα συμπεράσματα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι σήμερα θα έχω την ευκαιρία να μάθω περισσότερα σχετικά με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε αρκετές συναδέλφους που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να μιλήσουν. Πρώτα η κυρία Εστρέλα, η οποία είναι και η συγγήτρια της Επιτροπής όσον αφορά αυτό το θέμα με τη σχετική οδηγία. Ε, κυρία Εστρέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να καλωσορίσω την Υπουργό και να την ευχαριστήσω και για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε στην παρουσίασή της. Εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες προκειμένου να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, ώστε να συμφιλειωθεί η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή. αναμφισβήτητα ένας από τους τρόπους για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή τη συμφιλίωση είναι ε, να συμμεριζόμαστε τις οικογενειακές ευθύνες και η συμφιλίωση αυτή δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι και οι δύο. Κυρίως όσον αφορά στα οικογενειακά καθήκοντα. Να περάσω τώρα στα τη για την ε, άδεια μητρότητας. Δυστυχώς ε, δεν ήταν ε, αίσιο το τέλος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους ειδική Προεδρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και όχι μόνο εντός του Συμβουλίου, αυτό είναι γνωστό, αλλά ακόμα και εδώ στο Κοινοβούλιο. Στις συνεδριάσεις που έγιναν με τους κοιόδης εισηγητές ε, υπήρξε ευρεία συνένεση κυρίως ε, ως προς τα ουσιαστικά θέματα. Αλλά θα θέλαμε η συνένεση αυτή να διευρυνθεί ακόμα περαιτέρω διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους. Επιθυμία μας λοιπόν θα ήταν ακόμα και η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του ε, Κοινοβουλίου, το ΕΛΚ, να συμφωνήσει με τις βασικές προτάσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε αυτή την τόσο επιθυμητή συνένεση, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Η ερώτησή μου, κύριε Υφυπουργέ, είναι η εξή. Θεωρείτε ότι το Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει και με την πατρική άδεια στην οδηγία αυτή. Διότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δώσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία και να τους δείξουμε ότι οι ευθύνες πρέπει να είναι κοινέ και για τους δύο γονείς αν αφήσουμε εκτός οδηγίας ε, την άδεια πατρότητος, ουσιαστικά ε, εξαιρούμε τους άντρες από αυτή την ευθύνη. Και αυτό ε, είναι ένα πιστοδρομικό σήμα ε, επικίνδυνο και δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις θέσεις που πάντα υποστηρίζουμε εμείς. Και όταν λέω εμείς δεν αναφέρομαι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρομαι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Εμείς δηλαδή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Στρέλα. επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που είναι στα χέρια της Σουηδίας η Προεδρία και είναι κέρια σημασία στο να αναλάβετε ηγετικό ρόλο για αυτό το θέμα. Συμφωνώ επίσης απολύτως και με τη συνάδελφο κυρία Εστρέλα σε αυτά τα οποία ανέφερε. Το να συμπεριλάβουμε και την πατρική άδεια είναι σημαντικό Ξέρω ότι υπάρχει οδηγία για την ε, γονεϊκή άδεια, αλλά ξέρουμε ότι ακολουθεί μια πολύ αργή πορεία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση που γίνεται τώρα, σε αυτή την οδηγία, να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα. Υποστηρίζω λοιπόν την κυρία Στρέλα και θέλω και εγώ να ζητήσω το ίδιο από την Προεδρία. Και θα πρέπει και να συμπεριληφθεί και να υποστηριχθεί με οικονομικούς πόρους. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω αφορά τη χρονική περίοδο για την άδεια μητρότητα. Ξέρω ότι γίνεται μια σχετική συζήτηση γιατί κάποιε χώρε θέλουν μεγαλύτερη και κάποιε χώρε μικρότερη περίοδο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Το θέμα των 24 εβδομάδων που υποστηρίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Χρειαζόμαστε ε, μισό χρόνο για την γονεϊκή άδεια και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω ποια επιχειρήματα μπορεί να υπάρχουν, ποια επιχειρήματα θα μας απέτρεπαν από την πρόταση αυτή γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ο σωστός χρόνος για την άδεια μητρότητας. Επίσης, ε, ένα άλλο θέμα είναι οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες. Παρότι γνωρίζω ότι υπάρχει μια άλλη οδηγία που ασχολείται με αυτό το θέμα, έχω την εξής ερώτηση. Στην οδηγία αυτή υπάρχει κάποιο πεδίο για να μπει και αυτό το θέμα, για να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των γυναικών που είναι αυτοαπασχολούμενες και γυναικών που απασχολούνται από άλλους εργοδότες. Ευχαριστώ. Ε, Καλώς. Η κυρία Γκαρσία Πέρες το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Υπουργό για την παρουσία της εδώ και για το γεγονό ότι μα παρουσιάζει τι θέσει τη για ένα θέμα για το οποίο πιστεύω ότι η συνένεση είναι σαφή. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ε, στι λεπτομέρειε, αλλά ο βασικό στόχο που είναι να καταφέρουμε να συμφιλειώσουμε την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών στην ε, ε, εργασιακή του ζωή είναι θεμελιώδε. Γι' αυτό ακριβώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναζητήσει και μια κοινή θέση για το θέμα αυτό Ε, για την οδηγία την οποία συζητάμε. Θα ήθελα να παρουσιάσω την άποψή μου, ε, να πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι όσον αφορά στην πατρική άδεια. Αν θέλουμε πραγματικά να συμφιλιώσουμε την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, όπως είπε και η Εντίτ, δεν είναι μόνο οι γυναίκες αυτές που πρέπει να συμφιλιώσουν ε, τα δύο, ε, είναι οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια, ένα πιο ισότιμο εργασιακό πεδίο και να πάψουν να υπάρχουν οι ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις γυναίκες για να μπορούν να ανταγωνιστούν επίσης όρις στον εργασιακό βίο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Το να συμπεριληφθεί λοιπόν και η πατρική άδεια ανεξάρτητα από το τι ε, συμβαίνει είναι θεμελιώδες για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και το λέω αυτό θεμελιώδες διότι υπάρχουν κάποιες ε, ε, χώρες τις οποίες ε, ο άνδρας μπορεί να λάβει μέρος της γονεϊκής άδειας και ε, η άδεια αυτή αφορά στις γυναίκες και ο άνδρας μπορεί να πάρει τμήμα της άδειας. Αν θέλουμε να έχουμε ισότητα θα πρέπει να μιλάμε για δύο διαφορετικές άδειες που δεν θα μπορεί ο ένας να τη μεταφέρει ή να την εκχωρήσει στον άλλον. Η γυναίκα θα πρέπει να έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και στους πρώτους μήνες, τις πρώτες εβδομάδες ζωής του παιδιού της θα πρέπει οι άνδρες και οι γυναίκες να μπορούν να αναλάβουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα που σημαίνουν ε, να γίνει κάποιος γονιός, είτε άνδρας είτε γυναίκα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δίνουμε ένα πολύ στεναρό μήνυμα στο ότι ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όχι μόνο όσα λέμε επί χάρτου, αλλά θέλουμε πραγματικά να γίνουν ε, τμήμα της ζωής τους και η πατρική άδεια είναι θεμελιώδης για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστούμε για τις απόψεις σας. Δεν έχω κάποιο άλλο όνομα στον κατάλογο μιλητών. Οπότε στρέφουμε προς την καλεσμένη μας να μας κάνει κάποια σχόλια όσον αφορά τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το Συμβούλιο δεν έχει κάνει ακόμη συζήτηση σχετικά με την πατρική άδεια. Και είναι κάτι αυτό το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική οδηγία. Θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι οι απόψεις μας στη Σουηδία, αλλά σήμερα εδώ ο ρόλος μου είναι να εκπροσωπώ τα κράτη-μέλη από πλευράς της Προεδρίας και δεν έχουμε καν συζητήσει το θέμα αυτό ακόμη. Πάντως ευχαρίστω σημειώνω όλες τις απόψεις σας που μου αναφέρετε για το θέμα αυτό αυτό και για την κυρία Στέλλα και τον κύριο Ρουέδα και την κυρία Γκαρσία Περές. Ο κύριος Ρουέδα επίσης μίλησε και για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Ε, αυτό έχει ως στόχο την ε, άρση των ε, διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών που ασκούν μια ανεξάρτητη δραστηριότητα. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορές που παραμένουν στα κράτη-μέλη και κατά τις προσεχείς εβδομάδες οι προσπάθειές μας θα δείξουν πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάντως, ε, σαφώς ο στόχος μας ε, είναι γνωστός. Επίσης, ε, μας ρωτήσατε για τις 24 εβδομάδες. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν να παραταθεί η, μητρική, άδεια μητρότητας από 14 σε 18 εβδομάδες και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που συζητείται στο Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι αν θέλει κανείς να κάνει περαιτέρω σχόλια όσον αφορά τα μέλη της Επιτροπής εδώ. Αν όχι, αλλά τι βλέπω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να πω το καλώς όρισες κι εγώ στην Υπουργό να την ευχαριστήσω για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε και θα ήθελα να σας πω ότι εγώ είμαι συγγήτρια η γνωμοδότηση όσον αφορά αυτή την οδηγία ε, στα πλαίσια της Επιτροπής για τα κοινωνικά θέματα. Θα γίνει αύριο μια συνεδρίαση, αύριο το πρωί. Θα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψινου ε, ε, για αυτό το θέμα της οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εγώ υποστηρίζω ε, θερμά την ισότητα των ε, ευκαιριών και την κοινωνική ένταξη. Επιθυμώ πραγματικά να γίνει μια προσπάθεια προς τα μπρος όσον αφορά αυτό και να έχουμε, έχουμε μια, ε, ένα όραμα, μια εικόνα όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι εκπροσωπεί αυτό για τα παιδιά της θα πρέπει να δούμε πολιτικά μια λύση όσον αφορά το θέμα του διασμού επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Όλα αυτά αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό υποστηρίζω θερμά ότι σε αυτή την οδηγία υπάρχει δυνατότητα να εντάξουμε το θέμα που αφορά την πατρική άδεια. Τώρα, όσον αφορά την επέκταση για, το, την άδεια μητρότητα, θα ήθελα να πω ότι κατ' εμέ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια, τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γι' αυτό θα πρέπει πετύχουμε να πετύχουμε μια ε, ε, ε, αποτελεσματική άδεια μητρότητας η οποία να είναι προς όφελος του παιδιού. και για να υποστηρίξουμε αυτή την άδεια μητρότητας θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Υπουργό αν τώρα έχει υπάρξει μια οποιαδήποτε συζήτηση στο Συμβούλιο να έχουμε μια ε, έκθεση για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει ε, όσον αφορά τις πληρωμές, ε, τις μισούς μάλλον και πώς ακριβώς ισχύει το θέμα κατά τη διάρκεια την οποία κάποιος έχει άδεια μητρότητα. Σε ευχαριστώ, ε, Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και μας δώσατε τις άποψεις σας να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην Επιτροπή για τα κοινωνικά θέματα. Αλλά έχω και κάποιους άλλους ομιλήτριες. Πρώτα η κυρία Λούλινγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Υπουργό, διότι καθυστέρησα να έρθω στη συνεδρίαση για λόγους ε, ανεξαρτήτους της θελήσεώς μου και δυστυχώς δεν κατάφερα να ακούσω την ομιλία της Υπουργού. Είμαι συγγήτρια για την πρόταση οδηγίας που αφορά την μεταρρύθμιση της οδηγίας ε, ε, για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους συζύγους ε, που απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Ε, περίμενα πολλά από την Σουηδική Προεδρία, αλλά δεν έχουμε δει να συμβαίνουν πολλά και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τις προθέσεις σας. Η έκθεση εγκρίθηκε τον Απρίλιο. Έκανε κάποιες προσπάθειες και η Τσεχική Προεδρία αλλά είναι πια πολύ μεγάλη χρονική περίοδος που έχει μεσολαβήσει. Η έκθεσή μου εγκρίθηκε σχεδόν με ομοφωνία στο Κοινοβούλιο. Τώρα όσον αφορά την πρόταση που συζητάμε για την νέα οδηγία, για την γονεϊκή άδεια, ελπίζω ότι δεν θα εγκριθεί ως έχει, διότι για το πρόβλημα αυτό βλέπω ότι τείνουμε να διαπράξουμε τα ίδια σφάλματα που είχαμε διαπράξει όσον αφορά και την προστασία της μητρότητας. Δηλαδή προσπαθούμε να τα ανακατέψουμε όλα. Όταν είμαστε νομοθέτες με κοινή νομοθετική εξουσία πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Πρόκειται περί νομοθεσίας και όχι περί ενός καταλόγου με όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε να συμβούν. Μπορεί να είναι ευκταία όλα αυτά, αλλά εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να ασχοληθούμε με την νομοθεσία. Όταν έχουμε μεταρρύθμιση, όταν θέλουμε να επιτύχουμε μια μεταρρύθμιση της γονεϊκής άδειας, Χαιρόμαστε που και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε μέσα σε αυτή την οδηγία να τα βάλουμε όλα και πατρική άδεια και ίση αμοιβή και οτιδήποτε άλλο γιατί νομίζω ότι θα γελιοποιηθούμε έναντι της Επιτροπής και του Συμβουλίου με ένα τέτοιο ψήφισμα και υπάρχουν και μερικές τροπολογίες ακόμη χειρότερες. Εγώ θέλω να το πω ξεκάθαρα προς την Σουηδική Προεδρία γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή μας υπάρχουν ακόμη άτομα που ξέρουν πώς πρέπει να νομοθετούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Λούλινγκ. Η κυρία Ιλντα Φιγκουρέντο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όπως είπε η κυρία Λούλινγκ πριν από λίγο, υπάρχει, ε, βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πολύ αντίθετα προς από τη φορά που φανταζόμουν εγώ δεν πηγαίνουμε προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ισότητα, ίδιες ευκαιρίες, ίδια δικαιώματα για γυναίκες στο χώρο εργασίας, να εγγυηθούμε συγχρόνως ότι είναι σωματωμένες κοινωνικά και να εγγυηθούμε ότι μπορούν να έχουν ε, ε, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι έχουν δηλαδή αναλαμβάνουν τις ευθύνε του σαν μητέρε στη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει οι ίδιες τις ευκαιρίε στον χώρο εργασία. Θέματα μισθολογία. Υπάρχει το θέμα ότι οι, οι μητέρες και οι πατέρες θα πρέπει να ε, μοιράζονται τις ευθύνε στην οικογένεια, τι ευθύνε για τα παιδιά, τι υποχρώσεις του. Και το θέμα το να υπάρχει το δικαίωμα της ε, αδείας γονικής για τη μητέρα ή για τον πατέρα αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς να υπάρχουν συνέπειες για το εισόδημα της οικογένειας. Αυτά συνδέονται τα πράγματα. Θα πρέπει να τα δούμε συνολικά, να δούμε όλες αυτές τις πτυχές. Το να υποστηρίζουμε αρχές οι οποίες είναι ενδιαφέροντες αλλά αν δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα μέτρα, τι νόημα έχει. Χρειάζεται μια σωστή νομοθεσία η οποία διασφαλίζει αυτά τα δικαιώματα. Άρα, το ερώτημά μου προς την Υπουργό είναι το εξή. Η Προεδρία τι σκέφτεται να κάνει για να θέσουμε τέλος σε αυτό το χάσμα που υπάρχει. 30 χρόνια έχουν περάσει για αυτό το θέμα για να υπάρχει ισότητα μισολογική για τους άνδρες και τις γυναίκες. Και ποια μέτρα σκέφτεται η Προεδρία να λάβει για να δοθούν εγγυήσεις όσον αφορά την ε, επομισμό ευθυνών στην οικογενική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Πρόεδρος. Η κυρία Κώστα θα πάρει το λόγο τώρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ την Υφυπουργό κυρία Σόνεγκαρτ για την παρουσία της εδώ. Και νομίζω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προωθήσουμε την, ε, την όθεση που μας δίνεται λόγω της καθυστέρησης. Ε, κανονικά ήμασταν ε, μπροστά. Το 1994 όταν ε, έγινε η πρώτη οδηγία για την άδεια μητρότητας προχώρησαν τα πράγματα γιατί προχώρησε η νομοθεσία για πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα και την κρίση και την εργασιακή ε, κατάσταση των γυναικών και μέσω μιας μεγαλύτερης συμφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής ε, νομίζω ότι τα πράγματα θα μπορέσουν να προχωρήσουν ακόμα περαιτέρω. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτό το νέο βήμα γιατί είναι σημαντικό και ως μήνυμα. Η κυρία Λούλινγκ ε, επισήμανε ότι είμαστε νομοθέτες, το ξέρουμε όλοι και πρέπει να βρούμε και ένα σημείο ισορροπίας. Θα ήθελα να πω εδώ ότι θα ήταν σοβαρό να οπισθοχωρήσουμε σε σχέση με μια οδηγία η οποία έτυχε και μεγάλη συζήτηση και μεγάλη επεξεργασία στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει και μια προσμονή να προχωρήσουν τα πράγματα τόσο όσους συνυπευθυνότητα, δεν μπορούμε να δώσουμε σε καμία περίπτωση διαφορετικό μήνυμα, ε, όσο και συμβιβασμό την, ε, ε, της γονεϊκής άδειας και την αποζημίωση που δίνεται για την γονεϊκή άδεια και στους δύο γονείς. Το θέμα αυτό νομίζω συζητήθηκε και από την κυρία Εστρέλα. Και στην περίοδο αυτών των διάσημων τριών μηνών μετά τη γέννα, ο πατέρας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ε, πάρει άδεια, νομίζω ότι δεν μιλάμε για υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και πολιτικό μήνυμα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μιλάμε για υποχρεωτική άδεια του πατέρα ε, για τρεις μήνες. Εκεί νομίζω ήταν άλλωστε και το, το ακαθόδε σημείο. Αλλά μιλάμε για δικαίωμα του πατέρα σε αυτό το διάστημα να μπορεί να είναι και αυτός παρόν στα οικογενειακά ε, καθήκοντα. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και πολιτικό ζήτημα και ίσως και το Συμβούλιο, ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το υποστηρίξει και να το ενθαρρύνει για να μην σταματήσει και η συζήτηση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε και το θέμα των αυταποσχολούμενων εργαζομένων τόσο ανδρών όσο και γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κώστα. Η κυρία Μωρίν, το λόγο και μετά νομίζω ότι η καλεσμένη μας δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της. Θα μας δώσει όμως κάποια σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρέμβασή σας. Όλοι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Και δουλεύουμε τώρα πάνω σε αυτό το κείμενο που αφορά την άδεια μητρότητα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ε, διότι με την εξέλιξη της νομοθεσίας που προστατεύει τις γυναίκες μέσα στη μητρότητα, που προστατεύει τις γυναίκες ε, στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την απασχολησιμότητα των γυναικών. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει νομοθεσία που δεν θα συνοδεύεται ταυτόχρονα από διατάξεις που θα επιτρέπουν στις γυναίκες μέσα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να έχουν χώρους φύλαξης των παιδιών, παραδείγματος χάρη, παιδικούς σταθμούς, ε, ώστε να μπορούν να φέρνουν τα παιδιά τους κοντά στο χώρο εργασία του, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ζωτική σημασία για την εξισορρόπηση προσωπική και επαγγελματική ζωή. Και παράλληλα, δεν θα πρέπει να προβλέψουμε αύξηση ε, των αδειών μητρότητα χωρίς να προβλέψουμε και κάποια συνοδευτικά μέτρα ώστε να μπορούν να επανέλθουν στην ε, απασχόληση οι γυναίκες. Αυτό δεν το κάνουμε βέβαια μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον, το κάνουμε μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία προτείνουμε να είναι βιώσιμα. Η Astrid Λούλινγκ ε, μίλησε για ευχολόγια είναι δύσκολο το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και θέλουμε να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιο είναι το όραμα της Σουηδικής Προεδρίας για την έκθεση αυτή. Τι πιστεύετε ότι είναι δυνατόν και τι πιστεύετε ότι είναι εφικτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν και την κυρία Μωρίν. Θα πάρει το λόγο η καλεσμένη μας για σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι άκουσα διάφορες απόψεις. Όπως βλέπουμε, πολλά πράγματα θα πρέπει να προωθήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία στην οποία οι άνδρες και οι γυναίκες θα τη χάνουν ίσων ευκαιριών. Και νομίζω ότι αυτό επισημαίνει το γεγονός ότι ε, τα θέματα αυτά είναι δύσκολα, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικά συστήματα, τα οποία ε, ασχολούνται με την γονεϊκή άδεια, την άδεια μητρότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμφωλιώσουμε την οικογενειακή με την εργασιακή ζωή. Έχουμε διαφορετικούς τρόπους να εξετάζουμε τα θέματα και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Και θα πρέπει να επισημάνω ότι δεν υπάρχει θέση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη, όπως σας είπα στην αρχή, αλλά έχουμε διαπιστώσει πολλές αντιρρήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι διαφορετικά και χρειαζόμαστε χρόνο να συζητήσουμε αυτές τις διαφορές και να καταλήξουμε σε μία οδηγία η οποία θα έχει ε, χαρακτήρα εξελαχίστων. Θα πρέπει να το θυμόμαστε ότι η οδηγία αυτή είναι μια οδηγία εξελαχίστων που σημαίνει ότι θέτει τα κατώτερα δυνατά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πόσο διαφορετικές είναι οι χώρες μεταξύ τους και πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται τα θέματα αυτά. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα ε, με την παράταση της ε, άδεια μητρότητας και επίσης και το θέμα της υποχρεωτικής άδεια που ακούσαμε και προσφάτως είναι και αυτό πρόβλημα για κάποιες χώρες πολλές χώρες θεωρούν ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τουλάχιστον όχι τόσο διεξοδικά. Αυτά νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σας πω εν κατακλείδη. Θα πρέπει να θυμάμαστε ότι αυτή είναι μια οδηγία εξελαχίστων. Υπάρχουν χώρες με πολύ διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τις απόψεις του άλλου και θα πρέπει να βρούμε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παρουσιάσει προτάσεις, δεν είναι αρμοδιότητα της Προεδρίας αυτό και για την γονεϊκή άδεια οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που έχουν αναλάβει το καθήκον να ε, παρουσιάσουν μια οδηγία και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αποτελεί θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Με αυτά τα λόγια λοιπόν θα ήθελα να ολοκληρώσω τη συζήτηση από πλευρά μου για το θέμα της άδεια μητρότητα, αλλά θα ήθελα να πω λίγα πράγματα ακόμα για τους αυτοαποσχολούμενους. Έγινε κάποια ερώτηση σχετική. Η Σουηδική Προεδρία συνέχισε τις προσπάθειες της Τσεχικής Προεδρίας προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία στο ε, Συμβούλιο του Νοεμβρίου και αυτό είναι ο στόχος μας. και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες για διάφορα κράτη-μέλη και για το θέμα αυτό και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Στόχος όμως είναι να υπάρξει η πολιτική συμφωνία το Νοέμβριο. Να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, πρόσκληση να έρθω εδώ να σας ακούσω. Δυστυχώς πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την καλεσμένη μας για τις πληροφορίες που είχαμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι το θέμα είναι λίαν σημαντικό. Όλοι το έχουν καταλάβει. Πάλι σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία με τη συνέχεια της Προεδρίας και δι το να έχουμε μια καλή οδηγία για αυτό το σημαντικό θέμα. Γεια σας. discussion. Συνεχίζουμε με τη μερίσια διάταξη. Πριν να πάμε στο σημείο 5, χαρά να καλωσορίσω εγώ σήμερα μια, ένα, μια ομάδα από τη Σουηδία, επισκέπτες από το Γετεμπόρι και τα περίχωρα. Με γυναίκες που είναι στρατευμένες πραγματικά στο θέμα της ισότητας και ήρθαν εδώ να, ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν το, τη συνεδρίασή μας κατά το πρωινό και μετά να συζητήσουν αυτό το θέμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Σημείο 5. Στην ημερήσια διάταξη είναι το εξή. Το θέμα που αφορά πώς να υποστηρίξουμε την ισότητα συνδυάζοντας επαγγελματική ζωή με τα δικαιώματα ε, για την οικογένεια και την οικογενειακή ζώνη και είναι σαν συνέχεια της συζήτηση που είχαμε. Οι προϋποθέσεις για τη σημερινή συζήτηση είναι να έχουμε μια αρχική μικρή συζήτηση και μετά να ψηφίσουμε για το ψήφισμα. Το πλαίσιο αυτού του θέματος είναι ότι κάναμε σε ένα ερώτημα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ε, με αφορμή την συμφωνία για την ε, γονική άδεια το, κάτι το οποίο έχουν δεχθεί τα, οι κοινωνικοί εταίροι και τέλη του Νοεμβρίου θα, ληφθεί, θα εγκριθεί. Εμείς αποφασίσαμε στην Επιτροπή μας να κάνουμε προφορικές ερωτήσεις και να βγάλουμε αυτό το ψήφισμα και αυτό διότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μεγάλη σημασία η δική μας Επιτροπή και δι, δι Επιτροπή και, εν γέννη το Κοινοβούλιο να προσέξει στο να βελτιωθούν οι συνθήκες όσον, αφοράνε, όσον αφορούν το συνδυασμό επαγγελματική οικογενειακής ζωής. Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ισότητας. Ο βασικός στόχος του ψηφίσματος που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ε, όσον αφορά την γονική άδεια να δούμε διαφορετικούς τύπους οικογενειακών θα λέγαμε σχηματισμών διαφορετικούς τύπους οικογενειών και τι ακριβώς γίνεται με τις γονικές άδειες. Στο κείμενο ψηφίσματος προτείνεται βλέπουμε ότι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί είναι μια συμφωνία την οποία εμείς υποστηρίζουμε. Αλλά θέλουμε να δράξουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή τη συμφωνία σαν ένα πρώτο βήμα. Θέλουμε και άλλα μέτρα για να βελτιωθούν περαιτέρω οι δυνατότητες σε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά την ισότητα. Στο ψήφισμά μας κυρίως λαμβάνουμε, βλέπουμε το θέμα του, της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και θα λέγαμε είναι ένα, μια συμφωνία που εξασφαλίζει τα ελάχιστα και γι' αυτό το βλέπουμε σαν ένα πρώτο βήμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ε, αυτό συνδέεται με την παλιότερη συζήτηση που είχαμε για την πατρική άδεια. Έτσι για να δώσουμε ένα σίγμα ότι η ευθύνη για τα παιδιά δεν είναι μόνο για τη μητέρα αλλά και για τους πατέρες. Να δώσουμε λοιπόν σαφέστατο μήνυμα διότι φάνηκε ότι όταν έχουμε μια καλά συγκροτημένη γονική πατρική άδεια αυτό έχει θετικές συνέπειες. Έτσι υπάρχει μια καλύτερος καταμερισμός ανάμεσα στο μητέρα και το πατέρα και όταν ας πούμε έχει κανείς μια διαφυγή εισοδήματος αυτή γίνεται με ένα πιο δίκαιο τρόπο μέσω της ε, πατρικής αδείας και δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν επαγγελματική και κοινωνική ζωή παράλληλα. Και εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό. Αυτά σαν μια, ας το πούμε, μικρή εισήγηση για να σας διαγράψω το πλαίσιο όσον αφορά το ψήφισμα στο οποίο θα, θα ψηφίσουμε αργότερα. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκουρμάη. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο ήθελα να κάνω. Αλλά καθυστέρησα και γι' αυτό κράτησα το σχολείο μου για τώρα. Έχω δύο γιου, Ο μεγαλύτερο είναι 22 ετών και έμεινε τρει μήνε με τον πατέρα του στο σπίτι. Και αν δούμε την άποψη του παιδιού, υπάρχει τεράστια διαφορά γιατί δεν το είχαμε καταφέρει να μείνει και με το μικρότερο γιο. Πάντως ε, το παιδί χρειάζεται τον πατέρα του και ε, από την εμπειρία μου μετά από 22 χρόνια Πρέπει να σας το πω αυτό. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ του πατέρα και της μητέρας και πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε την ψαλίδα της διαφοράς αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, να μπορούν να εργάζονται και οι γυναίκες εφόσον χρειάζονται τα χρήματα για την οικογένεια. Και ήθελα να συνεισφέρω αυτή την προσωπική μου εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Ευχαριστούμε κύριε Αγκουμάη. Πολύ στη σημαντική η, η άποψή σας, δηλαδή να δούμε την, και την προπτική από, τη σκοπιά του παιδιού. Ευχαριστώ λοιπόν που μας σωθήξατε αυτό. Κύριε... Μάλιστα. Αναφέρατε στην εισαγωγή σας στο θέμα για το ψήφισμά σας είπατε θέματα τα οποία δεν ε, θίγονται στη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων. Θα πρέπει να προσέξουμε, να μην τα ανακατεύουμε όλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε την γονική, ε, ε, γονική άδεια, όχι την πατρική. Οι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται για την διαπραγμάτευση τη γονική. όταν θα καταλήξουν κάπου θα έρθουν ε, εδώ. Αλλά εμεί σε αυτή την οδηγία που αφορά τη γονική άδεια να μην ανεφέρουμε το θέμα της, ε, ζητάμε την πατρική άδεια. Θέματα ισότητας των μισθολογίας. Υπάρχει μια νομοθεσία από το 1975 όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τους μισθούς. Θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις χώρες μέλη. Είναι σωστές οι νομοθεσίες. Αν όμως οι χώρες και οι γυναίκες που πλήττονται δεν πάνε στα δικαστήρια, τι θέλετε να γίνει. Τους αφήνεις πόρτες ανοιχτές. Δεν αρκεί να κλαίγεται κανείς. Νομοθετική εργασία χρειάζεται δυνατή. Μπορούν να πούμε ακόμα ότι έχουμε τις διάφορες επιθυμίες και το ένα και το άλλο, αλλά ειλικρινά σας παρακαλώ μην τα ανακατεύουμε, τα μην τα κάνουμε αναχταρμά. Αν το κάνουμε θα, γίνουμε, θα γελιοποιηθούμε. Να πάει κανείς με μια, ένα τέτοιο ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Γιατί κάνετε, δημιουργείτε τέτοια κείμενα, πώς τα συντάξετε. η νομοθεσία πρέπει να είναι εφαρμόσιμη. Εμείς έχουμε, όταν έχουμε φέρει πίν δυνατότητα να, ε, να κάνουμε ένα έργο το οποίο είναι συν απόφαση, συν, να συνομοθετήσουμε καλώς. Αλλά όταν κάνουμε σε μια περίπτωση όπου κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία είναι διαφορετικό. Όταν έχουμε να κάνουμε θέματα στα οποία υπάρχει συναπόφαση, συνομοθεσία, θα πρέπει να είμαστε λογικοί, να μην τα ανακατεύουμε. Και τι τροπολογίε πραγματικά το είναι ακόμη πιο αστείε από το αρχικό κείμενο, ειλικρινά. Ευχαριστώ την κυρία Λούλιν. Έχω κι άλλε ομιλήτριε. Πρώτο όμω ο λόγο σε ένα ομιλητή. Μετά είναι η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Φιγκερέιντο, αλλά πρώτα ο Ραούλ θα πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Λούλινγκ, Εμείς εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είμαστε εθνικοί βουλευτές και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να διαμορφώσουμε νομοθετικές προτάσεις μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα όχι να αναζητήσουμε το ελάχιστο, αλλά να αναζητήσουμε το επιθυμητό μέγιστο για να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής του ε, λαού της Ευρώπης, όχι σε εθνικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν χώρες για τις οποίες θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα, στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αλλά εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθούμε με το γενικότερο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πώς θα τα προσαρμόσουν αυτά. Εδώ νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας να έχουμε μια εντελώς ευρωπαϊκή προοπτική. Επιστρέφω στα ισπανικά. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί κατανοώ απόλυτα ότι αυτό που προσπαθούμε να πούμε δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε με διαφορετικές πτυχές. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει πολλές διαστάσεις και το καθένα αποτελεί τμήμα του προβλήματος αλλά και της λύσης. Δεν μπορεί να μιλάμε για ισότητα και ίσες ευκαιρίες και για ισότητα δικαιωμάτων των γυναικών να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας αν δεν υπάρχει και η πτυχή της υποχρέωσης οι άνδρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους στον ιδιωτικό τομέα πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου μονομίσματος. Εάν τις διαχωρίσουμε δεν μιλάμε για ισότητα, μιλάμε για άλλο πράγμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα διαχωρίσουμε. Πρώτη σκέψη αυτή. Δεύτερη σκέψη. Φρονώνται όταν μιλάμε για μια οδηγία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι και φιλόδοξες για αυτό το στόχο και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι μα. Υπάρχει το ενδεχόμενο μετά από την εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη να έχουμε διαφορετικού ρυθμού προσέγγιση. Δεν λέω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, νομοθετικά είναι απαραίτητο. Αλλά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ευθύνη να χαράξουμε τον ορίζοντα. Και όχι να χαράξουμε έναν ορίζοντα ξεκινώντα από τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά ξεκινώντα από εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και ε, ε, δεν θα πρέπει να είμαστε στις πιο περιοριστικές νομοθεσίες αλλά θα πρέπει να είμαστε στις πιο προοδευτικές νομοθεσίες για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ως φάρος για τα υπόλοιπα. Αλλιώς δεν θα προχωρήσει η Ευρώπη, θα οπισθοχωρήσει. Είναι προφανέ ότι στο τέλος ε, το αποτέλεσμα θα είναι ένας μέσο όρο. αλλά ο μέσο όρο δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αν ξεκινάμε από έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Ας πάρουμε το ελάχιστο και τελεία. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ένα φιλόδοξο στόχο και με την συζήτηση που θα γίνει με τα κράτη-μέλη θα γίνει μια προσέγγιση που θα φτάνει πιο πολύ στο μέσο όρο, ε, και, αλλά δεν θα φτάσει στο ελάχιστο που φαίνεται να ζητούν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ραούλο Μέβα, σε ευχαριστούμε. Εγώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο για να διευκρινίσω κάτι. Όσον αφορά τη συμφωνία ε, ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους είναι σαφές για μας ότι είναι συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους όπου εμείς σαν κοινοβούλιο δεν μπορούμε να πειράσουμε τα πράγματα. Αντιθέτως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε με αυτό το ψήφισμα είναι να δείξουμε ότι εμείς είμαστε στρατευμένοι στο θέμα, έχουμε μια άποψη η οποία δείχνει ότι στο μέλλον στο έργο μας μπορούμε να προχωρήσουμε τις θέσεις μας όσον αφορά το θέμα τα ισοτήτων, ισότητα. Συγγνώμη. Δηλαδή ότι οι μητέρες και οι πατέρες να μπορούν να αναλάβουν από κοινού θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ευθύνη όσον αφορά τα παιδιά και είναι σημαντικό λοιπόν μέσω αυτού του ψηφίματος να δείξουμε ότι είναι ένα βήμα ε, εκ μέρους του Κοινοβουλίου. δεν είναι δεσμευτικό το ψήφισμα. Τώρα, ο λόγος στη κυρία Παπαδοπούλου και μετά η κυρία Φιγκερέιντα και μετά η κυρία Παβανόβα αλλά τώρα μέσω η κυρία Παπαδοπούλου. Α Ναι, ναι. Κάποιες. Πρόνοιες. Τις διατάξεις εννοεί. Συγγνώμη. Τις διατάξεις είναι πρόνοια. Πρόνοια. Οι θερμοπίδακες. Mm. Mm-hmm. αλλά δεν κατάλαβα καν που τρόπο τι είπε ο κάνει. Λέω είπε κάτι κυπριακό, άντε να το, να το μεταφράσει. Και ετοιμάζεται να πάρει και Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου. Η κυρία Φιγκερέιντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελέγχθησαν πολλά όσον αφορά αυτό το θέμα. Τώρα συζητάμε ένα ψήφισμα. Δεν είναι θέμα οδηγίας, νομοθεσίας. Ένα απλό ψήφισμα είναι όπου διατυπώνουμε την άποψη της Επιτροπή μας πάνω σε αυτήν την κατάσταση. Και εκφράζουμε την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά τις ίδιες ευκαιρίε, την ισότητα και τις δυνατότητες να συνδυάσουμε την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και δει τα δικαιώματα των μητέρων. Να υπάρχει μια εγγύηση. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν αξίζει να είμαστε, δεν αξίζει να υπάρχουμε σαν Επιτροπή. Είναι το καθήκον μας σαν Επιτροπή. Θα πρέπει να δράσουμε ούτω ώστε να κάνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται αυτές τις πτυχές. Ο στόχος ενό ψηφίσματο είναι να δημιουργήσει, να προκαλέσει την προσοχή του Συμβουλίου της Επιτροπής. Δεν μιλάμε για οδηγία. Η κυρία Λούλινγκ, λοιπόν, η συνάδελφός μας, νομίζω ότι δεν έχει καθόλου δίκιο σε αυτά που λέει. Πρόεδρος, ε, ε, σας ευχαριστώ κύριε Φιγκερέντο. Κύριε Πάβανόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου αλλά και την απογοήτευσή μου για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τη συζήτησή μας. Διότι εγώ ήρθα σε αυτή την επιτροπή, διότι από ό,τι είχα καταλάβει ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να μιλήσουμε για ισότητα των φύλων. Και οι εκλογείς, όλοι εκτός κοινοβουλίου, όλοι αναμένουν από εμά ότι θα προστατεύσουμε τις γυναίκες και θα μιλάμε υπέρ της ισότητας των φύλων. Δεν, θα, δεν είναι αντικείμενο της Επιτροπής μας η μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ε, οι επιχειρήσεις γενικά ή οι εργοδότες. Εμείς είμαστε Επιτροπή Γυναικών και μέσω της Επιτροπής μας έχουν την ευκαιρία να δουν να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Και όσοι πιστεύουν ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας ή δεν είναι αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε στην Επιτροπή μας, ε, μπορεί να πάει σε άλλη Επιτροπή, ας πάνε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, οπουδήποτε άλλο. Αλλά εμείς εδώ στην Επιτροπή μας αυτή τη δέσμευση αναλάβαμε, υποσχεθήκαμε, ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα δικαιώματα των γυναικών, όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, Μόλις επιστρέφω από την διάσκεψη EPCD στην Αιθιοπία και πρέπει να πω ότι ήταν απογοητευτικά τα, τα συμπεράσματα. Είδαμε ποια είναι η κατάσταση ε, των αναπτυσσομένων χωρών και πρέπει εμείς οι ανεπτυγμένες χώρες να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να τηρήσουν τους στόχους όσον αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής ε, των γυναικών και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Και όταν μιλάμε εδώ για την γονεϊκή άδεια, μας ενδιαφέρει να μιλάμε για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και υποστηρίζω στεναρά αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος, η κυρία Φιγκουερέιντο, να έχουμε κατά ότι μιλάμε για ένα ψήφισμα εδώ και μέσω αυτού του ψηφίσματος θα δείξουμε ότι έχει την αξιοπιστία η Επιτροπή μας ε, γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών. Και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στα, ε, στις προτεραιότητές μας και στους στόχους μας και να μην παρεκκλίνουμε από το βασικό στόχο για τον οποίο βρισκόμαστε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να δώσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στο κοινοβούλιο μας. Αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, στο μέλλον η Επιτροπή μας θα εξαφανιστεί. Δεν θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη θέσπιση νομοθεσίας. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να δίδουμε τη γνωμοδότησή μας για όλα τα θέματα νομοθεσίας από την πλευρά της τήρησης των δικαιωμάτων ε, ισότητας και προστασία των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Παβανόβα. Η κυρία Κράτσα έχει το λόγο. Πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αισθάνομαι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ε, ε, ε, ε I will, I will answer to my colleague, please, please, please. Θέλω να σας απαντήσω αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πιστεύω ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή ε, τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ρόλο της Επιτροπής μας. Αλλά θα ήθελα να επενθυμίσω, ίσως τα καινούργια μέλη χρειάζονται ιδιαίτερη υπενθύμηση, ότι εμείς είμαστε ένα πολιτικό σώμα και είμαστε μια κοινοβουλευτική επιτροπή και όχι μια μη κυβερνητική οργάνωση που υποστηρίζει μια θεματική και αυτός είναι ο στόχος της και το περιεχόμενό της. Έχουμε το λόμπι των γυναικών, το οποίο είναι αφοσιωμένο σε αυτό το ρόλο και είναι και για μας συμβουλευτικό όργανο. Έχουμε πολλές άλλες γυναικείες οργανώσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς είμαστε ένα πολιτικό σώμα που εργαζόμαστε για μια κοινωνία που θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη συνοχή και περισσότερες ευκαιρίες και δικαιοσύνη για τις γυναίκες. Και κάθε μας απόφαση πρέπει να εγγράφεται σε αυτό το, το γενικό στόχο. Κάθε κόμμα πολιτικό, κάθε ένας από εμά γιατί έχουμε την αυθύπαρτη προσωπικότητά μας και ευθύνη, καταγράφουμε με τις δικές μας απόψεις αυτό το στόχο. Αλλά δεν είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών, αν ένα πολιτικό σώμα και μια, ε, και και πολλές φορές με κοινοβουλευτική αρμοδιότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πιστεύω έστω και αν δεν είναι τώρα το περιεχόμενο και το πλαίσιο αυτής της συζήτησης πρέπει να τα υπενθυμίσουμε. ευχαριστώ. Uh, κυρία Κράτσα, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα είναι επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ. Επειδή ακριβώ είμαστε πολιτικό όργανο και ως Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να διευκρινίσουμε σαφώς ποιοι είναι οι ρόλοι μας και ποιες είναι οι διάφορες νομικές βάσεις που έχουμε σήμερα για να μπορέσουμε να λάβουμε δράση. Ένα παράδειγμα να σας κάνω. Έχουμε τρία θέματα να ε, συζητήσουμε. Το θέμα της συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την οδηγία για την άδεια μητρότητας, για την γονεϊκή άδεια. Έχουμε μία οδηγία την οποία συζητάμε από την προηγούμενη θητεία για το θέμα της διεύνησης της ε, άδειας μητρότητας και της πατρικής άδειας και έχουμε και μία πολύ σημαντική ε, πολιτική πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να λάβουμε μέσω ενός ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν τρεις διαφορετικούς χώρους έκφρασης είναι σαφές ότι θα υπάρχει μια έκθεση για την οδηγία, θα συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους και εμείς, θα ακούσουμε και την άποψή τους, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να παρέμβουμε αυτόνομα ως πολιτικό όργανο για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο ε, συμμερίζονται ευρύτατα οι Ευρωπαίες γυναίκες και ελπίζω και οι άνδρες. Ε, εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω. Η θέση της συναδέλφου Λούλινγκ φαίνεται να αναφέρεται στο γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να μπορέσουμε να εκφράσουμε την άποψή μας ή για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με αυτό ε, το αποτέλεσμα. Σαφώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό που συζητούν οι κοινωνικοί εταίροι, διότι πρόκειται για περίπλοκα θέματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό έγινε και το 1994 με την οδηγία για τη γονεϊκή άδεια. Σήμερα όμως υπάρχει μία νομική βάση, μία βάση νομιμότητας διαφορετική. Έχουμε τη συνθήκη και έχουμε περαιτέρω διαδικασίες, ε, χάρτα δικαιωμάτων. Και εκεί οι πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες είναι σε μια πολύ πιο προηγμένη βάση, πιο θεσμική βάση και επομένω εμεί έχουμε τη δυνατότητα και το καθήκον, όπω έλεγαν πριν κάποιοι συνάδελφοι, να εκφραστούμε αυτόνομα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε θέμα αυτό προ όλε τι κατευθύνσει και να συμφωνήσουμε με την ευρωπαϊκή κοινωνική γνώμη, να δούμε πού, σε τι φάση οριμότητας βρισκόμαστε και ως προς το Συμβούλιο, το είπα και πριν στην Υφοπουργό που ήταν εδώ και ε, ω προ του κοινωνικού εταίρου που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρόκειται για πολιτική πράξη. Δεν είναι μία πράξη μη κυβερνητική οργάνωση. Είμαστε μία επιτροπή που γνωρίζει το ρόλο τη και θέλει να επαναλάβει το ρόλο τη ε, στο πλαίσιο αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχε κάποια στιγμή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, το άκουσα αυτό, γιατί εγώ τότε ήμουν βουλευτή στην Ιταλία. Ε, πρόκειται για μια επιτροπή που ε, ασχολούνταν με όλα και με τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια κοινή αίσθηση και αυτό είναι να δώσουμε μια νέα όθηση στο ρόλο της Επιτροπής μας και θα πρέπει να συζητήσουμε την ουσία. Σαφώς μπορούμε να συζητήσουμε την ουσία ενός ψηφίσματος, αλλά το να πούμε ότι εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε πράγματα διότι θέλουμε να δώσουμε μια πολιτική κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι σοβαρό σε σχέση με το ρόλο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κώστα. Η κυρία Μπάουερ μετά η κυρία Νικολάη και να υπενθυμίσω ότι είχα γράψει στην ημερήσια διάτηξη ότι θα είχαμε ψηφοφορία 10 η ώρα, αλλά ότι θα προηγεί το μία συζήτηση γιατί δεν το πράξαμε νωρίτερα. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Και αμέσως μετά θα κάνουμε ψηφοφορία. Κυρία Μπάουερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω λίγε σύντομε παρατηρήσει για να συνεισφέρω κι εγώ στη συζήτηση. Έχω κι εγώ την εντύπωση ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε αργά ή γρήγορα. Ποιο είναι ο σημαντικό ρόλο τη Επιτροπή μα και ποια είναι ε, τα καθήκοντά μα. Αλλά και, ε, και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουμε. Πάντως κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε τα καθήκοντά μας. Ξέρω ότι είμαστε ένα πολιτικό όργανο, αλλά δεν είμαστε το Προεδρείο ενός κόμματος. Εδώ συζητάμε πολιτικές θέσεις. Είμαστε ένα νομοθετικό όργανο. Είμαστε ένα όργανο μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με νομοθετικά ζητήματα. Και είναι λογικό το να υπάρχει διάσταση απόψεων. Υπάρχουν διαφορές και στις λύσεις που προτείνονται. Υπάρχουν ε, νόμοι που υπάρχουν εδώ και 30 και 40 χρόνια, αλλά όταν οι νόμοι αυτοί δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί και δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν, όταν υπάρχει ένα θέμα για τις διαφορές αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η νομοθεσία, η σχετική νομοθεσία, γιατί υπάρχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το να μπορούμε να ανεβρίσκουμε λύσεις Θέλουμε να μπορούμε να προτείνουμε νομοθετικές προτάσεις και να έχουμε αποτελεσματική νομοθεσία. Δεν έχει κανένα νόημα τα πάντα να τα συμπεριλάβουμε σε ένα κείμενο να μιλάμε και για ε, δίκαιες αμοιβέ και για ε, πατρική άδεια. Δεν μπορούμε να συνδυάζουμε τα μέτρα προστασίας της εργασίας με άλλα θέματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία προτείνουμε δηλαδή τα νομοθετικά κείμενα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα οποία είναι αρμοδιότητά τους. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα βάλουμε μέσα σε ένα κείμενο. Έχουμε αρκετά νομοθετικά κείμενα, έχουμε αρκετές διατάξεις και σε νέε διατάξεις νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια, ε, όπως έχω εδώ το κατάλογο, είναι η κυρία Νικολάη. θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Ήδη είχαμε εφαρμογή τέτοιου συστήματος στη χώρα μου και λειτουργεί. Δε... Αν ήμασταν με κυβερνητική οργάνωση, ε, καταλαβαίνω, θα δρούσαμε διαφορετικά αλλά πολιτικά όταν δράει κανείς ότι σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες αρχές για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αλλιώς θα οργανώναμε διασκέψεις, ε, συνεδριάσεις, σεμινάρια. Θα θεωρώ ότι για μας είναι ότι είναι σημαντικό να δώσουμε το έμφαση στην κοινωνική ε, ένταξη, ενσωμάτωση των γυναικών, στις ίσες ευκαιρίες και να δούμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν ε, να αντιμετωπίσουμε και την υπάρχουσα κρίση. Εγώ θεωρώ για όλους αυτούς τους λόγους και με την ιδιότητα της, ε, και της πολιτικής μου ιδιότητα σαν φιλελεύθερη θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε. Ένα διαδικαστικό θέμα, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις επί της διαδικασίας την οποία ακολουθούμε. Η διαδικασία την οποία έχουμε είναι η εξή. Εδώ έχουμε μία πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που έχει ως αντικείμενο να εξετάσει τα νομικά ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία, την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις ε, οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων. Δεν έχουμε εδώ μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία σχετικά με την ε, γονεϊκή άδεια. Μπορεί να πούμε ότι είναι κρίμα που αυτό έχουμε ενώπιόν μας, αλλά αυτό που έχουμε είναι το ότι πρέπει να δώσουμε μια γνωμοδότηση για αυτή την ε, πρόταση οδηγίας. Αν νομίζετε ότι δεν είναι αρκετά καλή, πρέπει αρκετά καλό να το απορρίψουμε αλλά μια συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων είναι κάτι το οποίο ή μας βρίσκει σύμφωνος ή μας βρίσκει να διαφωνούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τις διαδικασίες αυτές είναι ότι μπορεί η Επιτροπή να μας προτείνει να εξετάσουμε την συμφωνία πλαίσιο παραδείγματος χάρη και αυτό είναι το σενάριο στο οποίο βρισκόμαστε και κανένα άλλο. Και αυτό ήθελα να διευκρινίσω για να μην μου καταλογίζετε διαφορετικές προθέσεις. Αν σας μιλήσω για τη γονική άδεια που έχουμε στο Λουξεμβούργο, έξι μήνες ε, με 1.500 ευρώ αποζημίωσης ε, μηνιαίως και μπορούν να πάρουν αυτήν άδεια στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και οι άνδρες και οι γυναίκες και αυτό νομίζω θα σας και σύμφωνου. Και αυτό εμείς το επιτύχαμε με την οδηγία την οποία θα καταργήσουμε και την οποία θα βελτιώσουμε τώρα. Τέσσερις μήνες είναι το ελάχιστο. Εμείς έχουμε έξι μήνες, 1500 ευρώ. Άρα μην νομίζετε ότι εγώ θέλω να καθυστερήσω οτιδήποτε. Εγώ ευχαρίστω θέλω να λέτε 6 μήνες και 1500 ευρώ μηνιαίως. Γιατί αυτό θα σήμαινε και ισότητα με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Επομένως, μην ε, με παρανοείτε αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά όταν έχουμε ψηφίσματα τα οποία θα μας γελιοποιήσουν ενώπιον του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ θέλω να μα προφυλάξω από αυτό. Και γι' αυτό έχουμε τις τροπολογίες μας τις οποίες θέλουμε να ψηφίσουμε. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Λούλινγκ. Πριν να κάνουμε ψηφοφορία, να διασαφηνίσουμε κάνα δύο πράγματα. Η συμφωνία που επιτεύχει ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους είναι κάτι στο οποίο το Κοινοβούλιο δεν έχει μπορεί να επηρεάσει τίποτα. Ίσως μόνο το Συμβούλιο θα μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Αυτό το οποίο τώρα θα ψηφίσουμε είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε ε, εδώ μπροστά μας για να συζητήσουμε με αφορμή τις ε, προφορικές ερωτήσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε οδηγία, νομοθεσία, ένα απλό ψήφισμα για να συζητήσουμε και να ε, πάρουμε ε, θέση, να θίξουμε κάποια θέματα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και είναι πραγματικά είναι πολύ ωραίο το ότι μπορούμε όλοι εδώ πέρα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Και είμαι πεπισμένη ότι όλοι εδώ οι συνάδελφοι, συναδέλφισες ε, σέβονται ότι κάποιος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από κάποιον άλλον. Όλες οι απόψεις γίνονται σεβαστές είναι ένα σωστό βήμα αυτό εδώ. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά ε, είναι ένα θέμα το πώς ακριβώς θεωρεί ο καθένας ότι θέλει να προχωρήσει στα θέματα της ισότητας. Με αυτόν τον τρόπο ας κλείσουμε το ε, διάλογο και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε 29 τροπολογίες προτείνω να πάρετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και θα προσπαθήσω να ψηφίσουμε θα λέω τα στα αγγλικά ο αναφερόμενος της θα χρησιμοποιήσω τα αγγλικά γιατί καμιά φορά δεν λειτουργεί καλά αν τώρα κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα να με ενημερώσει. Είσαστε έτοιμοι, έτοιμες όλοι, μπορούμε να προχωρήσουμε, αν όντως είναι όλα καλά. Λοιπόν, ψηφίζουμε τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε, βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Έχουμε 12 ψήφους υπέρ, 15 ψήφους κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Τροπολογία 23. Πρώτο τμήμα κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 23. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, Εννέα κατά και μία αποχή. Καταπίπτει η τροπολογία 22. Περνάμε στην τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπεριθμών 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, για την τροπολογία 3, την οποία παρουσίασα, για να μπορέσουμε ίσως να έχουμε μεγαλύτερη συνένεση εδώ στην Επιτροπή, θα ήθελα να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία, να διαγράψουμε δηλαδή το τμήμα τη τροπολογία εντό παρενθέσεων, να αφήσουμε δηλαδή μόνο τη διαρκώς μεγαλύτερη ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών και το υπόλοιπο το αποσύρω. Ε,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 Άρχεται η ψηφοφορία. The τη ψηφοφορία, Πέρας της ψηφοφορίας, 17 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Άρα ψηφίζουμε και το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7, ψήφι υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε. Για την τροπολογία 8 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, μία αποχή. Περνάμε στην πρώτη αιτιολογική σκέψη όπου έχουμε πέντε τμήματα. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ΣΥΦΙΠΕΡ. κατά, Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote closed. 10 ψήφοι υπέρ, 20 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι είναι δύσκολο να το δούμε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το τρίτο τμήμα. Πέρασε τη ψηφοφορία. 9 ψήφισαν υπέρ, 20 ψήφισαν κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Τέταρτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πέμπτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία no, it's not the final vote. It's... δεν είναι η τελική ψηφοφορία αυτή είναι για το πέμπτο τμήμα ψήφισαν όλοι Πέραση της ψηφοφορίας, 10 ψήφοι υπέρ, 16 ψήφοι κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. Τώρα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία, με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα με 17 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 13 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ όλους. Now we go to, uh, Yes, still Yes, because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 Eh, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο 6. Έχουμε περίπου 15 λεπτά πριν να δεχθούμε την επίσκεψη του Επιτρόπου Σπίτλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε προετοιμασίες εν ώψη ακροάσεων για τους ε, ε, υποδειχθέντες επιτρόπους. Λίγα πράγματα για τον κανονισμό που έχουμε όσον αφορά την εξέταση των υποδειχθέντων επιτρόπων. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω όλες τις συναδέλφισες ότι εσείς στα χαρτιά σας έχετε παράρτημα που περιγράφει το κανονιστικό πλαίσιο και πραγματικά σας προτρέπω όλες να το δείτε το οποίο αυτό το εγγραφό γιατί περιγράφει πώς ακριβώς γίνονται οι διαδικασίες αυτές. Οργανώνονται από κοινού, από τη διάσκεψη των Προέδρων και τους Προέδρους των Επιτρών, Επιτροπών. Ναι. Είχαμε λάβει μια, ένα χρονοδιάγραμμα από τη διάσκεψη των Προέδρων που λέει ότι οι ακροάσεις θα λάβουν χώρα την εβδομάδα 49 30 Νοεμβρίου, Δευτέρα με 4 Δεκεμβρίου και θα πρέπει θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και τη βδομάδα του Στραβούζου 25-26 Νοεμβρίου. Ε, θα μπορέσει ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε ότι έχουμε μικρό χρονικό διάστημα. Από το πότε ενημερωνόμαστε για το ποιοι έχουν προταθεί για, ε, για την Επιτροπή και αποφασίστηκε ότι οι ακροάσεις θα γίνουν ως εξής. Θα έχουμε πέντε κοινέ ερωτήσεις, οι ίδιες ερωτήσεις για όλους τους ε, πρωταθέντες. Και αυτές οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με τις ικανότητες, συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρωπαϊκής συνεργασίας, μια ανεξαρτησία προσωπική και ικανότητες, αρμοδιότητες της τομείς για τις οποίες έχουν προταθεί. Επίσης, ερωτήσεις για τις σχέσεις που έχουν με το Κοινοβούλιο και τις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Επίσης, ποιες είναι οι προτεραιότητες τους και γενικότερες πολιτικές ε, ερωτήσεις. Επιπλέον, η δυνατότητα που έχει κάθε επιτροπή είναι να προτείνει αν θέλουμε, αν θέλει η Επιτροπή, λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πέντε ερωτήσεις που θα αφορούν τον Επίτροπο τον οποίο έχει προταθεί. Σήμερα, στη σημερινή συνεδρίαση, θα έπρεπε να έχουμε μια συζήτηση. Ποιες ερωτήσεις μπορεί να είναι σχετικές από τη δική μας σκοπιά. Δεν θα λάβουμε απόφαση σήμερα, αλλά η συνάντηση των συντονιστών θα το αποφασίσει αργότερα. Να πω σύντομα απλώς κάποια πράγματα για κάποιες, θα το πούμε, προτάσεις. Και το κείμενο θα το δούνε εγγράφως όλοι οι συναδέλφισες, να γίνει σαφές δηλαδή. Μια μικρή ενημέρωση λοιπόν για κάποιες έτσι, πιθανές προτάσεις και στη συνέχεια θα χαρώ να έχω τις απόψεις σας πάνω σε αυτές. Μια ερώτηση θα μπορούσε να αφορά τη μελλοντική στρατηγική για τις ισότητες 2011-2015, τις νέες προκλήσεις. Ποιος είναι ένας, θα λέγαμε, οδικός χάρτης για την ε, ισότητα από το 2006-2010, μπορούμε να βρούμε καινούριε προκλήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γύρανση στον πληθυσμό, ότι αυτό το αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία μας. Θέματα ενσωμάτωσης στην κοινωνία, ολοκλήρωσης, μεταναστευτικά, Επίσης, πώς μπορούμε να δουλέψουμε συστηματικά για να εφαρμόσουμε το λεγόμενο gender mainstreaming στην νομοθεσία, αλλά και άλλες σημαντικοί και άλλες σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι. Επίσης το θέμα της οικονομικής ισότητας και της ανεξαρτησίας και όπως είπαμε νωρίτερα σήμερα, πώς θα μπορεί κανείς να συνδυάσει την επαγγελματική, την κοινωνική και την οικογενειακή ζωή. Τώρα, άλλη προτεραιότητά μας είναι πώς να προλάβουμε, πώς να μεταμετωπίσουμε και να εμποδίσουμε τη βία κατά των γενικών, την εμπορία ανθρώπων και πώς μπορούμε να βάλουμε, λάβουμε μέτρα τα οποία είναι προληπτικά και να υποστηρίξουμε αυτούς που είναι θύματα μιας τέτοιας αντιμετώπισης. Επίσης, το θέμα που έχει να κάνει με την κοινωνική ενσωμάτιση και τη μετανάστευση. Και κυρίως εδώ να δώσουμε έμφαση στα θέματα το, της ισότητας, δηλαδή με γυναίκες που είναι από άλλη, άλλης εθνικής καταγωγής και να διασφαλίσουμε και τα δικά τους δικαιώματα. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή για θέματα που θα μπορούσαν να είναι θέματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στους προταθέντες επιτρόπους. Το λόγο τώρα έχουν εδώ οι συναδέλφισες όσον αφορά αυτά τα θέματα που ανέφερα. Παρακαλώ, κυρία Γερόκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Και η παρατήρησή μου είναι σχετική. Έχω μια έκθεση για το θέμα, έχω κάνει μια έκθεση για τα δικαιώματα των Ρώμα και η Επιτροπή στον οδικό χάρτη της 2010 φύγει αυτά τα θέματα. Δεν έφτασε όμως αρκετά μακριά η Επιτροπή, δεν προχώρησε αρκετά. Το Κοινοβούλιο έχει διοθετήσει ψηφίσματα για τα δικαιώματα των Ρώμα και με ενδιαφέρει πολύ να θέσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα για τα δικαιώματα των Ρώμα και για την ένταξη των Ρώμα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το κατά πόσο ένας ε, υποψήφιος επίτροπος ε, έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, πόσο σημαντικό θεωρεί αυτό το θέμα από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης ε, και από πλευράς ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό θέμα για πολλά κράτη-μέλη και από δημογραφικής πλευράς υπάρχει το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού πολλές ε, δημογραφικές αλλαγές στον πληθυσμό των Ρώμα και υπάρχουν κράτη-μέλη όπου 40 έως 50% του ενεργού πληθυσμού έχουν ε, καταγωγή από τους Ρώμα. Με ενδιαφέρει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να ασκήσει πίεση για το θέμα αυτό και θέλουμε να έχουμε μια ομοιόμορφη πολιτική για τους Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι μα ενδιαφέρει η θέση ενό υποψηφίου επιτρόπου για το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δύο ερωτήματα έχω. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ε, σε τίνο στο χαρτοφυλάκιο θα ανήκει αυτή η Επιτροπή. Θα έχουμε κάποιο Επίτροπο για ανθρώπινα δικαιώματα ή θα είναι μια αρμοδιότητα που θα αφορά περισσότερο τον κοινωνικό τομέα, τις κοινωνικές υποθέσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πρώτα αυτό το θέμα του χαρτοφυλακίου για να ξέρουμε ε, σε ποιον θα απευθύνουμε τα ερωτήματά μας. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα, ζητώ συγγνώμη αν το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό το θέμα, όσον αφορά την ε, ψαλίδα της διαφορετικές αμοιβέ ε, ανδρών και γυναικών. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να θέσουμε μια τέτοια ερώτηση, διότι η δική μας Επιτροπή Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να συζητά τέτοια θέματα. Έχουμε ήδη μια έκθεση από πέρυσι για το θέμα αυτό. Και όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων, ε, δεν έχω σχετικό ερώτημα γιατί είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προφορική ερώτηση και δεν είναι βέβαιο αν ο επίτροπος αυτός θα έχει την αρμοδιότητα για το θέμα. Μπορεί κάποιος άλλος επίτροπος να είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό του εμπορίου ανθρώπων. Σήμερα ήδη το συζήτησα με κάποιον αρμόδιο από πλευράς Επιτροπής. Είναι ένα θέμα για το οποίο ήδη έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στο Συμβούλιο, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές ποιος επίτροπος θα έχει αυτή την αρμοδιότητα. Για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, ε, λοιπόν, είναι ένα ερώτημα που θεωρώ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε αν ε, αρμοδιότητα θα έχει ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για τις κοινωνικές υποθέσεις. Αλλά αυτό το ερώτημα είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα. Ε, Συμφωνώ με τις ερωτήσεις της Προέδρου και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα που έθεσε η κυρία Μπάουερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο σημαντικό θέμα του τι ακριβώς θέλει να κάνει η Ευρώπη για την πολιτική συνεργασία, κυρίως όσον αφορά στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται ε, σε αυτό που συμβαίνει για παράδειγμα στην Αφρική, την ενδυνάμωση των γυναικών στις ε, τρίτες χώρες και φυσικά και τη μεγαλύτερη συμμετοχή ε, τους ε, Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με πιο στεναρή παρουσία των γυναικών σε αυτή την κατάσταση. Κυρία Κονέλησεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλη μου την καρδιά με την πρόταση της κυρίας Μπάουερ να ρωτήσουμε για το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μας τη δουλειά και επίσης να διασφαλίσουμε ότι αν ε, συγκεράσουμε τα θέματα της ισότητας των φύλων με τα θέματα απασχόλησης θα υπάρχει εξορθολογισμός όλων των θεμάτων που άπτονται των ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς των εργασιών τη ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα το διασφαλίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε και κάποια θέματα για την χρηματοοικονομική κρίση. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η νέα επιτροπή που συστάθηκε για τα θέματα αυτά ασχολείται με τα θέματα της ισότητας των φύλων στα πλαίσια των εργασιών τους και θα πρέπει να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό. Επιπλέον, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, να καθορίσουμε συγκεκριμένα πράγματα για την επόμενη πενταετία. Επί το ψήφισμα που μόλις υιοθετήσαμε, η άδεια πατρότητας, αν δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην οδηγία που προτείνεται αυτή τη στιγμή, η Κομισιόν θα προτείνει μια οδηγία για την άδεια πατρότητας, διότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να υπάρχει. Να πιέσουμε λοιπόν αυτόν ή αυτήν που θα έρθει για την ε, ε, ακρόαση για το θέμα αυτό. Κάτι ακόμα σημαντικό είναι κατά πόσο ο νέος Επίτροπος θα είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση για χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν την οδηγία ίσης μεταχείρισης. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να προσπαθήσουμε να εκμεεύσουμε κάποιες συγκεκριμένες υποσχέσεις για την επόμενη πενταετία που θα υποχρεώσουμε ε, τον μελλοντικό Επίτροπο να τηρήσει. Ευχαριστώ κυρία Κονέλη. Ήταν και όλες τις συναδέλφες για σημαντικές παρατηρήσεις. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεως στη συνεδρία συντονιστών. Υπάρχουν κάποια θέματα που έθεσε η κυρία Μπάουερ και ισχύουν ακόμη. Θα ζητήσω λοιπόν από τη Γραμματεία να κοιτάξουν το θέμα του κανονιστικού πλαισίου, να είναι σαφής για να έχουμε απαντήσει τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Μπάουερ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε βάσει των, ε, τη σύσταση της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο για όλους τους Επιτρόπους. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο θα αναλάβει ποιο χαρτοφυλάκιο και αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι γνωστό όταν η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για τις προτεραιότητες. Γι' αυτό ακριβώς και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών πρότεινε και η διάσκεψη των Προέδρων συμφώνησε σε αυτό να επισυνάψει σε αυτό το γενικό ερωτηματολόγιο ένα παράρτημα το οποίο θα περιλαμβάνει τις προτεραιότητες με ένα μέγιστο πέντε προτεραιοτήτων που θα έχουν υποδείξει όλες οι επιτροπές. Οι επίτροποι θα απαντήσουν γραπτός σε αυτό το ερωτηματολόγιο που σημαίνει ότι κάθε επίτροπος θα απαντήσει γραπτός και στο τμήμα του παραρτήματος που θα άπτεται των αρμοδιοτήτων του ή της. Και έτσι θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατανομή των χαρτοφυλακίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι όλοι τώρα βλέπουν ποιες είναι οι προποθέσεις. Να αφήσουμε λοιπόν το θέμα εδώ να το αφήσουμε στους συντονιστές για να λάβουν απόφαση το απόγευμα. Και πριν. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι η επίσκεψη του. Από τον Επίτροπο κ. Σπίντλα Είναι εδώ απ' έξω. Μάλλον τον καλωσορίζουμε τώρα. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά... Με μεγάλη χαρά επαναλαμβάνω, χαιρετώ τον Επίτροπο κύριο Σπίτλα ε, εδώ στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Επίτροπος ε, είναι υπεύθυνο για θέματα κοινωνικά, απασχόληση και ίσες ευκαιρίες. Και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι η γενική εικόνα του Επιτρόπου για το τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας σε θέματα ισότητας. Και ένα σημαντικό θέμα νομίζω που υποστηρίζουν ε, και οι συναδέλφοι εδώ και θα θέλαμε περαιτέρω ενημέρωση είναι το θέμα ε, της ισότητας ε, για την περίοδο 2006-2010 και επίσης για το Ινστιτούτο για θέματα ισότητας και μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Χαιρόμαστε λοιπόν που είσαστε εδώ παρόν μαζί μας κύριε Επίτροπη και θα πάρετε αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, χαίρομαι ιδιαίτερως που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σβένσον για την πρόσκλησή της. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, το θέμα της ισότητας των φίλων και των δικαιωμάτων των γυναικών ήταν στο κέντρο των ενασχολήσεών μου. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το 2004. Πριν από πέντε χρόνια το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είχε αύξηση 2,5% ενώ σήμερα η ανάπτυξη βρίσκεται σε κάμψη και το ΑΕΠ της Ένωσης ε, φέτος ε, μειώνεται κατά 4%. Η τρέχουσα κρίση που δεν είχε προηγούμενο μετά τον, ε, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια κρίση που δημιουργεί τεράστιες ζημίες όσον αφορά την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούλιο του 2009 η ανεργία ήταν 9,5% του ενεργού πληθυσμού και η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία θα αυξηθεί και θα φτάσει το 11% στα τέλη του 2010. Όπως γνωρίζετε, οι πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας συνήθως είναι αυτές που πρώτες πλήττονται από την κρίση. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης επί της ισότητας ανδρών και γυναικών. Όμως, η ανάλυση της εξέλιξης των ποσοστών ανεργίας από το Μάιο του 2008 δείχνει ότι οι άνδρες επλήγησαν περισσότερο από ότι οι γυναίκες από την ανεργία. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει να έχουμε ίδια ποσοστά ανεργίας. Αυτό εξηγείται από το ότι οι τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, ήταν οι τομείς που απασχολούν περισσότερο άνδρες, δηλαδή οι κατασκευές και η βιομηχανία. Όμως αυτή η τάση μειώνεται τους τελευταίους μήνες. Η ανεργία των ανδρών και των γυναικών αυξάνεται με την ίδια ταχύτητα τώρα πια. Και αυτό με οδηγεί σε τρεις διαπιστώσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες πλήττονται εξίσου από την κρίση. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις της κρίσης επί της ισότητας ανδρών και γυναικών και να τονίσουμε τη σημασία των πολιτικών ισότητας που μπορούν να αποτελέσουν μια στρατηγική για την έξοδο από την κρίση. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα τα οποία εξαγάγαμε από την Υπουργική Διάσκεψη που οργάνωσε η Σουηδική Προεδρία στις 15 και 16 Οκτωβρίου του 2009. Η κρίση τονίζει την αναγκαιότητα του να δώσουμε έμφαση στις πολιτικές ισότητας. Αφενός μεν η κρίση δεν πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για να χάσουμε τα κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών, αφετέρου δε η κρίση μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε συμπεριφορές και να προωθήσουμε τις πολιτικές ισότητας ε, όσον αφορά τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, τα τελευταία πέντε χρόνια η Επιτροπή ανέπτυξε δράσεις υπέρ της ισότητας γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πολιτικός άξονας αφενός ήταν ο ένας και ο νομοθετικός άξονας ήταν ο δεύτερος. Και οι δύο άξονες είναι βεβαίως συμπληρωματικοί. Όπως γνωρίζετε, η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι κάτι το οποίο έχει συμπεριληφθεί στις συνθήκες από το 1957. Η ισότητα των φύλων λοιπόν αποτελεί μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια απαραίτητη συνθήκη για την υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και αν η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε σημαντικές προόδους, γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την τρέχουσα κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να ανανεώσουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ισότητα των φύλων και ο χάρτης πορείας για την ισότητα ανδρών και γυναικών για την περίοδο 2006-2010 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006 ακριβώς εκφράζει αυτή τη δέσμευση της Επιτροπής. Στο πλαίσιο τη της αυτού του χάρτη πορεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και θα ήθελα να αναφέρω τρεις από αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις για να καταπολεμήσουμε τη διαφορά στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η διαφορά στην αμοιβή που είναι 17% αυτή τη στιγμή είναι απολύτως απαράδεκτη. Οι λόγοι για αυτή τη διαφορά είναι πολλοί. Καταρχήν το ότι εμένει μια άμεση διάκριση έναντι των γυναικών. Δεύτερον, ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να πλήττονται από τα στερεότυπα και δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε ορισμένους τομείς. Και τρίτον, οι γυναίκες είναι θύματα διαχωρισμού στην αγορά εργασίας και συχνά οι γυναίκες περιορίζονται σε τομείς ή σε επαγγέλματα που έχουν μικρότερη αξία ή στους οποίους απολαμβάνουν μικρότερη αμοιβή. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι το Μάρτιο ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίηση για να κινητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ξεκινώντα από του κοινωνικού εταίρους, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώ αυτή τη διαφορά στην αμοιβή. Η εκστρατεία αυτή ήταν πολύ επιτυχημένη και η Επιτροπή θέλει να την παρατείνει και το 2010. Ακόμη τονίσαμε ότι είναι σημαντική η καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην οικονομική και πολιτική ζωή. Προσφάτως έχουν υλοποιηθεί πρόοδοι και είναι πολύ θετικό ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή το ποσοστό γυναικών είναι το πιο υψηλό, είναι 35%. Όμως, συνεχίζουν να είναι απαραίτητες ε, έντονες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, όπου οι γυναίκες εκπροσωπούν μόνο το 24% στα εθνικά κοινοβούλια. Όπως επίσης και στις επιχειρήσεις, όπου οι γυναίκες εκπροσωπούν λιγότερο από 11% των μελών διοικητικών συμβουλίων που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τον Ιούνιο του 2008, δημιουργήσαμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τις γυναίκες σε θέσεις ε, λήψης αποφάσεων. Το 2009 επίσης ορίστηκαν πολλά άτομα, διορίστηκαν σε σημαντικές θέσεις στην, ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο ενδιαφέρεται ιδιαίτερω για την εκπροσώπηση των γυναικών στην Επιτροπή. Μια τρίτη σημαντική πρωτοβουλία τη Επιτροπή είναι η δημιουργία του Ινστιτούτου των Φίλων στο Βίλνιου. Γνωρίζω πόσο πολύ και εσεί ενδιαφέρεστε για αυτό το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να λειτουργήσει και μπορεί να ξεκινήσει τι δραστηριότητε του άμεσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου θα εγκρίνει το πρώτο του πρόγραμμα εργασιών, το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων δημιουργείται αυτή τη στιγμή και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όρισε δύο γυναίκες εκπροσώπους στο φόρουμ αυτό. Η διευθύντρια του Ινστιτούτου και το προσωπικό της, το οποίο τώρα προσλαμβάνεται, θα εγκατασταθούν ε, στο Βίλνιου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου πολύ σύντομα. Γνωρίζω ότι είναι πολλές οι προσδοκίες από αυτό το Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Υπόστηριξη το Ινστιτούτο ώστε να μπορέσει να επιτύχει. Κυρίε και κύριοι, εκτό από την πολιτική διάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει και την κοινοτική νομοθεσία σε θέματα ισότητα ανδρών και γυναικών. Το 2006, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν την κωδικοποιημένη οδηγία που περιλαμβάνει σε ένα και μόνο κείμενο πολλές οδηγίες που αφορούν την ίση μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ισότητα των Φύλων είναι πλέον περισσότερο κατανοητή και καλύτερα ευανάγνωστη από τους Ευρωπαίους πολίτες και ταυτόχρονα βελτιώθηκε και ενισχύθηκε η σχετική νομοθεσία. Τον Οκτώβριο του 2008 εγκρίθηκε το πακέτο για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής και σίγουρα αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων. Όπως γνωρίζετε, αυτό το πακέτο αποτελείται από τρεις μείζονες πρωτοβουλίες. Πρώτον, μια νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Δεύτερον, μια δεύτερη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση των συζύγων που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και τρίτον μια έκθεση για την υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνας για θέματα υποδομών φύλαξης παιδιών. Επίσης, πρέπει να αναφέρω στο ίδιο πλαίσιο τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά τη γονεϊκή άδεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση οδηγίας τον Ιούλιο του 2009 με στόχο την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας στα κράτη-μέλη. Φρονώ ότι μπορούμε όλοι να χαιρετήσουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία ενισχύει τα δικαιώματα που έχουν σχέση με τη γονεϊκή άδεια. Επανέρχομαι στις δύο νομοθετικές προτάσεις που υπάρχουν επιτάπητος. Γνωρίζω και συμμερίζομαι το μεγάλο σας ενδιαφέρον για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών σε θέματα άδεια μητρότητας. Όπως γνωρίζετε και όπως ακούσατε και σήμερα το πρωί, το Συμβούλιο έχει υποβάλει πολλές επιφυλάξεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας, συνεχίζοντας να έχουμε υψηλέ φιλοδοξίες. Καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωστοποιήσει τη θέση του στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή και από τα δύο θεσμικά όργανα. Επίσης, συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τονίζει τη σημασία που έχει το να επιτρέψουμε στους πατέρες να παίξουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα από τις υπηρεσίε μου να κάνουν μια μελέτη για το κόστος και τα ωφέλη μιας ενδεχόμενης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό τον τομέα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα. Όπως γνωρίζετε, αυτή η πρόταση αποσκοπεί κυρίως στο να προσφέρει στους συζύγους που εργάζονται σε οικογενικές επιχειρήσεις να έχουν ίσο επίπεδο προστασίας, τουλάχιστον ίσο με το επίπεδο προστασίας που προσφέρεται στους αυτοαπασχολούμενους. Επίσης, να προσφέρει στις γυναίκες που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα τη δυνατότητα του να υποφελούνται, αν το επιθυμούν, από άδεια μητρότητα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι οι Υπουργοί θα υιοθετήσουν μια κοινή θέση στο Συμβούλιο της 30 Νοεμβρίου. Επ' αυτής της θα μπορέσει να καταστεί δυνατή μια σύντομη, μια γρήγορη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το δρόμο τον οποίο έχουμε διασχίσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Σίγουρα αυτέ οι πρόοδοι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν χωρί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερω τη δική σα Επιτροπή. Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω την κυρία Ζαμπόρσκα, η οποία προείδρευσε με μεγάλη επιτυχία την Επιτροπή σας κατά την προηγούμενη θητεία. Είχαμε υποδειγματική συνεργασία. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχηθώ, κυρία Σβένσον, κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Ε, δεν θα είναι εύκολος ο ρόλος σας μέσα στην τρέχουσα συγκυρία και βλέποντας τις προκλήσεις που υπάρχουν στα θέματα ισότητας των φύλων μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος ανέφερε στο πολιτικό του πρόγραμμα για την επόμενη θητεία της Επιτροπής ότι θα είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ισότητα των φύλων. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να ερμηνευθεί με δύο σημαντικές πρωτοβουλίες υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα ανδρών και γυναικών οι υπηρεσίες μου διεξάγουν μία διεξοδική ανάλυση επιπτώσεων και χωρίς να προδικάσω το περιεχόμενο του νέου πλαισίου, νομίζω ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες πριν από πέντε χρόνια, δυστυχώς πρέπει να πω, είναι τα ίδια. Έξι τομείς προτεραιότητας υπάρχουν στο χάρτη πορείας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί κατά τη γνώμη μου. Όμως η οικονομική κρίση μας υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε το να οπισθοδρομήσουμε στα θέματα δικαιωμάτων των γυναικών. Εξάλλου, η δημιουργία νέων προκλήσεων, όπως είναι η δημογραφική γύρανση, η αλλαγή του κλίματος ή η μετανάστευση, μας υποχρεώνουν να υλοποιήσουμε νέες πολιτικές. Σας καλώ λοιπόν να συνεισφέρετε ενεργά στην προετοιμασία αυτού του νέου στρατηγικού πλαισίου και θέλω να προσπαθήσουμε να βρούμε και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Επίσης, στην αρχή της επόμενης χρονιάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τη νέα της πρόταση για τη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση μετά το 2010. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα αυτής της στρατηγικής. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα η δική σας Επιτροπή να συνεργαστεί στενά στην προετοιμασία αυτής της νέας στρατηγικής. Τέλος, το 2010 θα είναι επίσης το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2010 θα πρέπει να καταδείξουν το πρόβλημα της φτώχειας των γυναικών και να επιτρέψουν να βρεθούν μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, επιτρέψατε μου κλείνοντα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά τη σημασία που έχει η ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο μέσα από μια ισχυρή εταιρική σχέση και μέσα από ένα ανοιχτό διάλογο θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερες πρόοδους στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Σπίτλα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που είχαμε για το ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, για την περίοδο των 5 ετών. Επίσης, εκ μέρους της Επιτροπής μας να ευχαριστήσω και για τη συνεργασία που είχαμε κατά την προηγούμενη θητεία και είμαι πεπισμένη ότι πραγματικά ότι εδώ στην Επιτροπή όλοι οι συναδέλφοι σας έχουμε τις φιλοδοξίες μας και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχουν γίνει πολλά κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια και ξέρουμε ότι όμως πολλά πρέπει να γίνουν και θα συνεργαστούμε και φυσικά να ενισχύσουμε όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, στα, όσον αφορά την ισότητα. Και πραγματικά ε, περιμένουμε πώς και πώς τη συνεργασία, τη μελλοντική και διάλογο για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Έχω μια σειρά όμως συναδελφισών που θέλουν να θέσουν ενδεχομένω ερωτήματα και πρώτη στην Ιγκουμάη είναι στον κατάλογο μιλητό η κυρία Μπάουερ μετά, η κυρία Τόμσεν επίση, η κυρία Κράτσα φυσικά και η κυρία Γερόκα. Καταρχήν, στην κυρία Γκουμάη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι τυχερή γιατί μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σας ε, κατά την προηγούμενη θητεία και θεωρώ ότι ο Επίτροπός μας και η ομάδα του έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά σε θέματα ισότητας των φύλων. Σκα δεν είναι τυχαίο, διότι ο κύριος Μπαρόσο προσπάθησε να βάλει πολύ ψηλά την ατζέντα σε θέματα ισότητας των φύλων και θεωρώ ότι όλοι οι επίτροποι το θεώρησαν δεδομένο ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάτι λιγότερο του 30% να σε γυναίκες. Είναι κρίμα που φεύγουν πολλές γυναίκες επίτροποι και δεν έρχονται νέες γυναίκες για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Εγώ πρότεινα για, από κάθε κυβέρνηση να προτείνεται ένας άντρας και μία γυναίκα ε, για τη θέση του Επιτρόπου και από εκεί και πέρα να επιλέγετε αυτόν που είναι καλύτερος για τη θέση. Ο κύριο Μπαρόζο όταν ένας επίτροπος δεν ήταν αρκετά καλός για μάσος ω κοινοβούλιο χρειάστηκε να πληρώσει υψηλό τίμημα. Ε, θα πρέπει να κατανοούν ότι οι γυναίκες είναι το 52% όχι μόνο ω φυσική παρουσία αλλά και στην εξουσία. Ε, μιλήσατε για τον οδικό χάρτη της ισότητας των φύλων. Ε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εξαντλούνται, φτάνουμε στο 2010 σχεδόν Επομένως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική για την επόμενη πενταετία. Ε, ο Επίτροπος φυσικά που θα αναλάβει τα, ο του κυρίου Σπίτλαρ πρέπει να είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, διότι θεωρώ ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι προεξάρχον. Συζητήσατε και για την ε, διάσκεψη του Πεκίνου και το θέμα είναι πού θα ε, βρισκόμαστε τώρα. Ε, να δούμε και τι ακριβώς γίνεται. Εξαρτάται και από την τσεχική κυβέρνηση το θέμα. ευτυχώς ο κύριος Κλάους υπέγραψε χθες τη συνθήκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθεια και εγώ ως ιστορικό ε, ξέρω ότι όταν μιλάει για τα διατάγματα είναι το ίδιο σαν να μιλάει και για την ε, συνθήκη του Βάλκλαφ ε, και εγώ πρέπει να σας πω ότι απογοητεύτηκα ιδιαίτερα διότι η δήλωση δεν θα φτάσει στους πολίτες, διότι η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους τσέχους πολίτες. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Όπως οι Βρετανοί όμως και οι Πολωνοί ζήτησαν ε, να μην συμπεριληφθούν στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι Τσέχοι θα μπορούσαν να το είχαν κάνει νωρίτερα, ήταν άλλος όμως ο Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος βέβαια ήταν ο ίδιος και τότε. Λίγα σχόλια για αυτά που είπατε. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την έναρξη της κρίσης, ε, το, ζήσαμε το πρώτο κύμα, ε, υπάρχει όμως και το δεύτερο κύμα το οποίο αφορά περισσότερο τις γυναίκες διότι ε, απασχολούνται περισσότερο σε θέσεις μερικής απασχόλησης και οι περισσότερες έχουν επισφαλή συμβόλαια. Το 2007 είχαμε το έτος ε, για την ισότητα των φύλων και εκεί νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό κείμενο. Ε, όλη τη χρονιά είχαμε εργασίες και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Και ε, τότε θυμάμαι ότι το χάσμα ήταν μόνο 15% και οι γυναίκες έπρεπε να εργαστούν περισσότερες μέρες, ε, αλλά όταν κοιτάξαμε τα στατιστικά πέρσι διαπιστώσαμε ότι το χάσμα των πληρωμών της μισθοδεσίας είναι ανώτερο του 15%. Και οι γυναίκε πρέπει να πιέσουν ιδιαίτερα για να λάβουν, τις ίδιες να την ίδια μισθοδοσία. Χαίρομαι ιδιαίτερα, είχαμε μια εξαιρετική έκθεση, αλλά αν όντω είναι έτσι τα πράγματα, χρειαζόμαστε άλλα 70 χρόνια για να κλείσει αυτό το χάσμα των πληρωμών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και φυσικά δεν ε, πρέπει να περιμένουμε 70 χρόνια. Τώρα, για την επόμενη χρονιά, ε, είπατε ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ένδυας αλλά αυτό έχει και ένα γυναικείο πρόσωπο και θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο. Όσον αφορά τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματική ζωής ε, είναι γεγονό ότι τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι δημογραφικέ αλλαγέ, όπω ε, είπατε κι εσεί, και η οικογένεια με τον παραδοσιακή τη μορφή δεν υπάρχει πλέον, οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τι νέε μορφέ οικογένεια. Μία ερώτηση. Έχετε πληροφορίε από τον κύριο Μπαρόζο σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει με το χαρτοφυλάκιο για τις γυναίκες επιτρόπους και για τα πιο καυτά θέματα, αν θέλετε. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με τον τρόπο που ανοίξατε εσείς ε, για τα θέματα της ζώτας των φίλων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας δουλειά. Δεν είστε κάποιος που απλά ασχολείστε με τα θέματα αυτά, αλλά είστε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα και επειδή είστε πατέρας που έμεινε σπίτι για τα παιδιά του, όπως είπα σήμερα ε, το πρωί στη συνεδρίαση, ο άντρα μου είχε την εξαιρετική ευκαιρία να μπορέσει να μείνει σπίτι με τα παιδιά του και είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να μπορεί να έχει και τον πατέρα του και τη μητέρα του στο σπίτι. Αν λοιπόν μπορέσουμε να το μάθουμε από την πρώτη του ηλικία ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν και τον πατέρα του και τον πατέρα του και είναι ίσοι, ε, θα ήταν εξαιρετικό. Σα συγχαίρω λοιπόν για άλλη μια φορά για τη δουλειά σα και είμαστε πολύ τυχεροί και για την πρόεδρο που έχουμε γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ω πρόεδρο. Ευχαριστώ την κυρία Γκουμάη. Κυρία Μπάουερ, μετά κυρία Τόμσεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Γκουρμάη. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το ότι ήρθατε εδώ και είναι σημαντικό να καταγράψουμε αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί και αυτά τα οποία ακόμη απομένουν να κάνουμε. Διότι αρκετά σημεία εκκρεμούν και πρέπει να επιτευχθούν. Είπατε κι εσείς ότι οι προτεραιότητες για τη μελλοντική στρατηγική παραμένουν οι ίδιες. Όχι γιατί δεν καταφέραμε να επινοήσουμε κάτι νέο, αλλά διότι δεν έχουν επιληθεί ακόμη τα προβλήματα. Είναι αρκετά σημαντικά αυτά τα θέματα και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τέξεις. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα ενώπιόν μας, το θέμα της άδειας μητρότητας. Και γνωρίζετε ότι είναι ένα θέμα που διχάζει το κοινοβουλίο μας. Όχι διότι αμφιβάλλουμε ε, ε, για το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και πατρική άδεια, αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το αν μπορούμε ε, κάτω από τον τίτλο της υγείας και ασφάλειας να μπει και αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είχατε υποβάλει μια πρόταση για το θέμα της πατρικής άδειας. Και πιστεύω ότι είναι πολύ προτιμότερο να το έχουμε σαν χωριστό θέμα παρά να το αναμειγνύουμε με το θέμα της υγείας και ασφάλειας. Υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας για τις γυναίκες. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι αυτή, αν έχετε κάποιο σχετικό σχέδιο, αν ε, το έχετε δρομολογήσει, αν περιμένετε κάποιο μήνυμα από το Κοινοβούλιο, ποιες είναι οι προθέσεις σας. Και μετά από αυτά που είπατε κι εσείς και αυτά που είπε και η κυρία Γκουρμάη, επειδή έχουμε πολλούς νόμους σε αυτό το τομέα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας. Θα χρειαστεί να περιμένουμε 70 χρόνια ή 100 χρόνια για να φτάσουμε να έχουμε τελικά ίση αμοιβή για ίση εργασία. τα δικαστήρια αργούν πάρα πολύ στα θέματα αυτά και η νομοθεσία κατά της διακριτικής μεταχείρισης θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ίσες συνθήκες. Υπάρχουν νομοθετικά κείμενα τα οποία πρέπει να αναθεωρήσουμε Πρέπει να ενισχύσουμε τα νομοθετικά όργανα Διαφορετικά, για να αλλάξουν αυτά τα προβλήματα, για να αλλάξουν αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια παραμένοντας τα ίδια προβλήματα. Θα εξετάσετε λοιπόν το θέμα της επιβολής της νομοθεσίας όσον αφορά αυτό το θέμα. Και έχω και άλλη μια ερώτηση. Αν μπορείτε, θα ήθελα να μας πληροφορήσετε για τις εξελίξεις ε, σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των επιτρόπων. Θα υπάρχει κάποιος επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες ε, ισότητα των φύλων θα είναι στη δική του αρμοδιότητα ή θα παραμείνει η τωρινή κατανομή αρμοδιοτήτων. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μπάουρ. Κυρία Τόμψεν, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσετε για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας σε σχέση με την κρίση ε, και κυρίω λαμβάνοντα υπόψη την πτυχή τη ισότητα των φέλων. Όπως είπατε κι εσείς, στην αρχή πλήχθηκαν οι άνδρες ε, από την κρίση στον οικοδομικό τομέα, στον ε, τομέα των μεταφορών και ούτω καθεξής και τώρα διαπιστώνουμε ότι η ανεργία αρχίζει να πλήττει στο ίδιο επίπεδο και τους άνδρες και τις γυναίκες. Αλλά τι θα γίνει στο μέλλον, διότι εξ όσων διαπιστώνω εγώ, με χαμηλότερο φορολογικό εισόδημα ε, οι απελήσεις έχουν αρχίσει να αυξάνονται ε, ακόμα και στο δημόσιο τομέα και οι απολύσεις είναι κυρίως των γυναίκες. Στο μέλλον λοιπόν θα διαπιστώσουμε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες άνεργες από ότι άνδρες. Όλες οι κυβερνήσεις στην ε, Ευρώπη όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να καταπολεμήσουν την ανεργία. Αυτό που έγινε χθε ήταν ότι εγώ ήμουν μιλήτρια σε ένα μεγάλο διεθνές ε, συνέδριο στη Δανία για την ε, ενεργειακή απόδοση και όλοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι όταν παρουσίασε, παρουσίασα το πρόγραμμα για την ε, ενεργειακή απόδοση και από εκεί και πέρα έχουμε και πάρα πολλές σχετικές επενδύσεις. αλλά αυτή τη στιγμή το 80% των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα είναι άνδρες. Θα διασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο όλοι μας ότι όλα όσα επενδύονται από τα θεσμικά όργανα θα ασχολούνται και με το θέμα της ισότητας των φύλων ώστε να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης για τις γυναίκες. Διότι όταν το είπα αυτό στις σκηνές, ε, στο κοινό συγγνώμη χθε, διαπίστωσα ότι δεν το ήξεραν το πρόβλημα ε, και ε, είπαν ότι πρέπει να προάγουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τις γυναίκες. Η καταπολέμηση λοιπόν της κρίσης μέσω επενδύσεων πώς λαμβάνει υπόψη της το θέμα ισότητας των φύλων. Δεύτερον, το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ναι, κάθε μέρα λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τη Δανία. Πότε θα έχει η Δανία το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, διότι η Δανία ακόμα δεν έχει σχετικό Ινστιτούτο. Εστάλει μια επιστολή ε, στη Δανία το Μάρτιο του 2007 και δεν έχει συμβεί τίποτα έκτοτε. Ανησυχεί ο κόσμος, απαιτεί Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αν ένας από τους τέσσερις νέους ηγέτες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν και από τη χώρα σας και καλό θα ήταν είστε υπέρ του να είναι γυναίκα στην Ιρλανδία όλοι όσοι ψήφισαν κατά των ε, γυναικών ουσιαστικά ε, πρέπει να γίνει κάτι γιατί έχουν βαρεθεί όλοι να βλέπουν άντρες με κουστούμια στις θέσεις ε, τις υπεύθυνε. Θα πρέπει να έχουμε και γυναίκες να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γερόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα επιτέγματά σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείξατε τα τελευταία πέντε χρόνια και γιατί δώσατε υψηλή προτεραιότητα στο θέμα των Ρώμα. Χαίρομαι ιδιαίτερως ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε το θέμα των Ρώμα και το ότι είναι οικονομικό θέμα το να συμπεριλαμβάνονται και οι Ρώμα στην ε, ε, οικονομική δραστηριότητα και στο εργατικό δυναμικό. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Αναφέρατε το χάρτη πορείας και στις προτεραιότητες έχει αναφερθεί ε, το θέμα της διαφοράς αμοιβών και σημαντικό είναι και το θέμα των γυναικών Ρωμά. Υπάρχουν και άλλα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους Ρωμά και ε, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτά, αλλά οι εξελίξεις στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι πραγματικά κάτι συμβαίνει. Τώρα, για το μέλλον θα ήθελα να σας ρωτήσω εφόσον το 2010 θα θεσπιστούν και τα νέα μέτρα, η νέα στρατηγική της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Η κινητοποίηση των φτωχότερων στρωμάτων είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα προωθήσει η Επιτροπή. Και τι θα κάνει σχετικά με την ε, ε, συμπερίληψη και των φτωχότερων στρωμάτων στην οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, Ποια είναι η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα των Ρώμα. Για τα υπάρχοντα εργαλεία, τι γνώμη έχετε για την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε παραδείγματο χάρη και θα υπάρξει και κάποιο νομικό μέσο ε, για τα επόμενα χρόνια. Θα το θεωρούσα πολύ σημαντικό εγώ. Επίσης, για την νέα επιτροπή, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας ε, Ποιος θα έπρεπε να έχει το αρμόδιο χαρτοφυλάκιο. Τα τελευταία πέντε χρόνια εσείς αναλάβατε δεσμεύσεις και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει ότι είναι ένα σημαντικό θέμα θα μπορούσατε να μας πείτε αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σχετικά και αν θα είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλώς. Η κυρία Νίλσεν τώρα. Ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τον απολογισμό που έκανα. Ε, υπεγραμμίζεται την κρίση που μας έχει πλήξει εδώ και ένα χρόνο. Ε, επίσης, ε, υπάρχει το θέμα της ανισότητας των, ε, της μισολογίας ε, ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά απ' την άλλη αυτή η οδηγία που υπάρχει από το 1975 και είναι κρίμα λοιπόν που δεν έχει αναθεωρηθεί έκτοτε και τώρα είναι πήγον. Ελέγχθη εξάλλου ότι τα, οι συνθήκες είναι αρνητικές, χειροτερεύουν και οι ανισότητες γίνονται όλο και πιο επώδυνες λυπάμαι που δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Δεύτερο τώρα, και το αυτό δεν θα είναι επίση θετικό, μας αφορά, μας, είπατε, μα υποσχεθήκατε μια οδηγία για το θέμα που έχει να κάνει με τη συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακή ζωής. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτό το θέμα δεν το έχετε δει το θέμα που έχει να κάνει με την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή είναι πολύ σημαντικό, όπως και η ε, μερική απασχόληση, η ευελιξία, η μητρική άδεια, η πατρική, όλα αυτά τα θέματα μας αφορούν και έχουν συνέπειες, μίζωνες, ε, σημασία συνέπειες στη ζωή των γυναικών. Θα ήταν καλό να μας δώσετε μια απάντηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Και τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Παπαδοπούλου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν και εγώ θα συγχαρώ τον κύριο Σπίλτα για τη γόνιμη συνεισφορά του στα θέματα απασχόληση κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών. Να κάνω μια ερώτηση εκ μέρου τη κυρία Κράτσα, η οποία ζήτησε συγγνώμη και ήθελα να την υποβάλει την ερώτηση και είναι η ακόλουθη μετά από την πλούσια πολιτική καριέρα, κύριε Σπίλτα, που είχετε και μάλιστα με ευαισθησία όσον αφορά την ισορροπία των ρόλων των δύο φύλων και κυρίως μετά από πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρμοδιότητα την προώθηση του ρόλου των γυναικών, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που εμποδίζει την αντιμετώπιση της ανισότητας σε όλα τα επίπεδα, στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της πολιτικής, στον ιδιωτικό χώρο παρόλη την πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί από παντού παρόλε τις πολιτικές εκστρατεία ενημέρωση, χρηματοδοτήσει, νομοθεσία τα πράγματα προχωρούν μεν αλλά με αργά βήματα. ποιο είναι το βασικό ε, συμπέρασμα που έχετε εσεί για αυτήν την καθυστέρηση. Αυτή ήταν η ερώτηση τη κυρία Κράτσα και είναι συναφή και με τη δική μου ερώτηση. Και εγώ έχω διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόοδο στα θέματα ισότητας γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά υπάρχουν σοβαρά δημοκρατικά ελλείμματα. Το πρώτο είναι το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άντρε και γυναίκες και οι άνισες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και το δεύτερο είναι οι άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η οικονομική κρίση, συμφωνώ μαζί σας κύριε Σπίλτα, ότι πλήττει τις πολιτικές ισότητας ε, η ανεργία πλήττει τις γυναίκες, η φτώχεια πλήττει τις γυναίκες και η μείωση των θέσεων εργασίας οπωσδήποτε θα πλήξει τις γυναίκες στο εγγύς μέλλον. Η ερώτηση μου είναι ξεκάθαρη. Πρώτον, ποια δραστικά μέτρα θα μπορούσε να υιοθετήσει μια κυβέρνηση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε πιο άμεσα αποτελέσματα και επιτάχυση. Θεωρώ ότι το gender budgeting είναι ένα δραστικό μέτρο να αποφασίσουν δηλαδή οι διάφορες εθνικές κυβερνήσεις όταν καταρτίζουν προϋπολογισμούς να διοχετεύουν συγκεκριμένα κονδύλια σε συγκεκριμένες πολιτικές ισότητας. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε επί Γερμανικής Προεδρίας, θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματική και είναι ένας τομέας όπου μπορεί πράγματι να έχουμε αποτελέσματα, στον gender parity. Και η δεύτερη ερώτηση μου αφορά τις επιλογές που θα έχει ο κύριος Μπαρόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός ίσως να ξαναμπεί η ποσόστοση ώστε να γνωρίζουμε ότι κάθε εθνική κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να βάλει υποψήφιους άνδρες και γυναίκες και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα να υπάρχει ένας προκαθορισμένος αριθμός γυναικών έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που δεν πετυχαίνουμε με άλλες πολιτικές. Δηλαδή θέλουμε δραστικές αποφάσεις και μέτρα. Η ποσόστοση κατά την άποψή μου και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα δραστικό μέτρο για να έχουμε περισσότερες γυναίκες commissioners, επιτρόπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδοπούλου. Πολλές, πολλές ερωτήσεις για τον Επίτροπο. Για να δούμε, ο κύριος Σπίτλε θα προσπαθήσει να μας δώσει απαντήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ε, στη σειρά που τις άκουσα τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. ποια είναι η κατάσταση με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Θα ήθελα να πω η κατάσταση είναι ανοιχτή. Ο, χθες ο πρόεδρος υπέγραψε επικύρωση της συνθήκη. Τώρα ξέρουμε ποια είναι η νομική βάση και γίνεται και μπορούμε να πούμε τώρα ξεκίνησε η εργασία για την ε, κατανομή των χαρτοφυλικίων. Οι πληροφορίες που έχω εγώ δεν είναι τόσο σαφείς για να μπορέσω να κάνω δηλώσεις ε, άμεσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής σίγουρα προσπαθεί να πετύχει ώστε να τον περισσότερες θέσεις για γυναίκες. Και είναι και επίσης σαφές ε, οι χώρες μέλη ε, δεν αντιδρούν. Ε, αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει τώρα. Τώρα η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων είναι ανοιχτή. Θεωρώ μπορούμε να έχουμε κάποια ιδέα με την παρέμβαση του Προέδρου στο Κοινοβούλιο πριν από την, τον ορισμό του και σίγουρα θα υπάρξουν κάποια χαρτοφυκλάκια για τα δικαιώματα του ανθρώπου, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όλα τα άλλα θέματα είναι ανοιχτά. Τώρα, αν ήταν να πω κάτι για πιο συγκεκριμένα πράγματα για το μέλλον αυτής της πολιτικής θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε μια φάση πολύ ευαίσθητη. Έχουμε με τη διατύπωση ε, ε, εγγράφων σημαντικά, στρατηγικής φύσεως και όπως εγώ προσπάθησα να είμαι σαφή στην εισαγωγή μου λέγοντας ότι θέλω να συνεργαστώ στενά μαζί σας για να προετοιμάσω αυτό το στρατηγικό έγγραφο διότι όπως έχουν και να έχουν τα πράγματα, μέχρι τον Ιανουάριο θα είμαι επίτροπος. Με, το, σε καλύτερο μέρος της εργασίας, το πιο σημαντικό θα γίνει αυτό το χρονικό διάστημα και γι' αυτό να σας πω ότι είμαι ε, διατεθειμένος να δω την ουσία και να συνεργαστώ μαζί σας και να ενισχύσουμε την ιδέα ε, σε όλα τα έγγραφα στρατηγικής βίσεως την πτυχή για την ισότητα των ε, φύλων για να μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο να βγούμε από την ε, κρίση. Η κυρία Μπάουερ τώρα για τα ε, μητρική άδεια, τη γονική άδεια. Ξέρετε ότι εγώ είμαι υπέρ της γονικής άδειας για πολλούς λόγους και λόγω της εμπειρίας της προσωπικής μου δηλαδή αλλά Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι πάντα, είμαστε σε μια κατάσταση που είναι ευαίσθητη και περίπλοκη. Οπότε τι το ερώτημα. Η νομική βάση μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε σε αυτή την οδηγία και το θέμα της ε, πατρικής άδειας. Κατ' περιπλέκονται τα πράγματα. Αν υπάρξει μια δυναμική, ε, αλλά δεν το πιστεύω εγώ ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πρόοδο. Και το θέμα που τίθεται πάντοτε είναι ότι θέλουμε ουσιαστική πρόοδο. Αν, θέλουμε να, αν καταλήξουμε αυτή την οδηγή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει μια άλλη οδηγία. Έχουμε συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και έχουμε ζητήσει να δουν και το θέμα της πατρικής άδειας. Δεν πήραν θέση οι κοινωνικοί εταίροι, οπότε σημαίνει η Επιτροπή έχει τα χέρια ελεύθερα παραμένει στη δική μου στρατηγική και όπως έχουν τα πράγματα τώρα έχουμε χώρο να προχωρήσουμε. Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οι ουσιαστικές φυσικά. Τώρα, η εφαρμογή των δικαιωμάτων είναι ένα θέμα συζήτησης που είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες που έχουμε στα χέρια μας για να ενισχύσουμε, να επιβάλλουμε το δίκαιο Και πραγματικά εμεί μπορούμε να απαιτήσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο μια δήλωση. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε. Είναι θέμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε πολύ. Όσον αφορά τώρα για την οδηγία για κατά των διακρίσεων, έχουμε ξεκινήσει 14 ε, διαδικασίες για παραβάσεις που έχουν γίνει, 17 συγγνώμη, και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας. Και είναι κάτι το οποίο ε, αφορά εμένα και είναι ανάμεσα στις διαδικασίες που προχωρώ. Είναι ένα θέμα λοιπόν πάνω στο οποίο δουλεύουμε και χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, ένα μέσο είναι ότι έχουμε, έχουμε χρησιμοποιήσει, δημιουργήσει ένα οργανισμό για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτό που αφορά τους φορείς ισότητας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ενίσχυση σε αυτό το έργο και σε μεθόδους που μπορούν να είναι πιο χρήσιμες σε σχέση με το σήμερα. Κατ' εμέ λοιπόν η οδηγία για τιμής χρήση σε σχέση με το θέμα που έχει να κάνει με τις φορείς ισότητας θα πρέπει να ενισχύσει την προστασία της ιδέας ε, για την ισότητα και τη μη διάκριση, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στην Ευρώπη για να ενισχύσουμε τη ε, θέση των φορέων ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η κυρία Τόμσεν. Για ε, αυτά που είπαμε με την ανεργία, έθιξε αυτό το θέμα. εμείς είχαμε την ιδέα ότι η ισότητα των ευκαιριών είναι ένας τρόπος για να βγούμε από την κρίση. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όλα τα μέλη της κοινωνίας σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή σε όλες μας τις δράσεις, σε όλες τις αλλαγές που κάνουμε, να κοιτάμε την πτυχή που έχει να κάνει με τα φύλλα. Καλά υπογραμμίσατε πολύ σαφέστατα. Καλύτερα από ό,τι είχα σκεφτεί εγώ, αλλά υπάρχει η ιδέα η πολιτική να περάσουμε σε άλλες μεθόδους μπορούν να μας οδηγήσει σε αλλαγές όπου έχουμε να κάνουμε μια νέα κατάσταση όπου μπορεί να δει κανείς το θέμα της απασχόλησης ανθρώπων και γυναικών και περνώντα στις μελλοντικέ μας δράσεις να εντάξουμε αυτή τη στρατηγική και πρέπει συνεχώς να βλέπουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν την ισότητα διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ή δε μη μπορούν να χειροτερεύσουν. Η στρατηγική μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλο τον δυνασμό που είναι παρόν για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα, για το θέμα που έχει να κάνει με το, τη διαφορές στις μισολογικές. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει μια ιδέα η οποία ίσως να μην ξεκινά από την Επιτροπή, αλλά την ενίσχυσε η Επιτροπή σε αυτή την προηγούμενη πενταετία ε, νομοθετικά για πολλούς λόγους. Η πρώτη αιτία είναι με αυτόν τον τρόπο ε, υπογραμμίζοντας την κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική ακόμα στη σημερινή κοινωνία και σε μια κοινωνία όπου έχουμε στοιχεία μπορεί να δείξει κανείς πραγματικά τι μεγάλες διαφορές στις μισθολογικές Γι' αυτό λοιπόν δράσαμε έτσι. Κάτι άλλο είναι αν μειωθεί αυτό το χάσμα, βελτιώνεται η θέση των γυναικών. Με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Επίσης, υπογραμμίσατε για το θέμα για μια νέα οδηγία κάνοντας μελέτες, βλέποντας το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις μελέτες, λοιπόν, δεν είναι ικανοποιητικά και δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να βελτιώσει την νομοθεσία. Επιπλέον, οι συζητήσεις με τις κοινωνικούς εταίρους έδωσε αποτελέσματα, θα έλεγα, κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά, φτωχά. Θα δουλέψουμε ως πάνω σε αυτό και δεν αποκλείω και τη δυνατότητα να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο. Η κυρία Γιώργα τώρα. Αναφέρθηκε για τους Ρώμα, μειονότητες. Δεν ξέρω αν οι, αξιολο... οι εκτιμήσεις είναι σωστές. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι εμείς την προηγούμενη θητεία ε, αυτό το θέμα το κοιτάξαμε και φυσικά σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο ή μάλλον περισσότερο το Κοινοβούλιο ήταν πιο έντονο. Ε, κάναμε μια προσπάθεια και βλέπει κανείς ότι είναι ένα θέμα πλέον ευρωπαϊκής διαστάσεως και κοιτάμε να δούμε ποια είναι τα μέσα που μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά από αυτές τις πολιτικές που ασκούμε σήμερα δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτού του θέματος συγκεκριμένα, διότι είναι ευαίσθητο θέμα, υπάρχουν αντιφάσεις και ισορροπίες πολύ λεπτές. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε ε, τις διαδοχές προεδρίες, αγγλική και σπανική, για να βρούμε μια λύση. Διότι έχουμε ήδη έχουμε συλλέξει αρκετή εμπειρία και έχουμε να κάνουμε πλέον με προεδρίες οι οποίες για πολλούς και διάφορους λόγους είναι, τους είναι σε αυτό το θέμα και αυτή θα ήταν η δυνατότητα κατ' εμέ για να δημιουργήσουμε μια δυναμική για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το θέμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους Ρώμα ειλικρινά θεωρώ ότι ε, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προεριώσουμε μόνο στη βάση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Είναι πιο ευρύ, πιο, πολύ πιο ευρύ αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με την ενημέρωση, την κοινωνική διάσταση κατ' εμέ θα ήταν καλό να λάβουμε υπόψη την εξής ιδέα, ότι ορισμένοι επίτροποι ενδεχομένω να έχουν ε, μεγαλύτερο βάρος από ό,τι κάποιοι άλλοι. Για μένα όμως είναι ένα θέμα αυτό που λέμε mainstream δεν είναι κάτι που περιφραγωγίζεται σε συγκεκριμένα μόνο ε, χρωτοφυλάκια. Η κυρία Παπαδοπούλου τώρα. Και η κυρία Κράτσα. Μου θέσανε ουσιαστικά ερωτήματα. Για ποιους λόγους τώρα, ποιες είναι οι αιτίες. Κατ' εμέ, είναι η παράδοση ανακλονισμοί. δεν έχει καταλάβει κανείς ενδεχομένως ότι οι κοινωνίες έχουν εξελιχθεί, έχουν, μεγαλώσει, έχουν προχωρήσει. Υπάρχει ο παραδοσιακός, η παράδοση. Φυσικά, συζητώντας, μπορείς κανείς να επιτεθεί και στις παραδόσεις, οι οποίες είναι, λειτουργούν αντιδραστικά. Κατ' για την αποτελεσματικότητα είναι η ενημέρωση, να μην περιορίζονται οι γυναίκες σε ένα περιορισμένο τομέα ε, ενημέρωσης κατάρτισης. Έχουμε και το Ινστιτούτο στη Βαρκελώνα, ε, Βαρκελώνας. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια ανάπτυξη, να δημιουργηθούν υποδομές και το άλλο θέμα που προκύπτει είναι το θέμα της εξουσίας. Δεν μπορεί να πει κανείς φυσικά να περάσει εξουσία όλες στις γυναίκες, αλλά τουλάχιστον η μισή. Το θέμα αυτό της ποσόστοσης τώρα για την Επιτροπή είναι μια ιδέα η οποία είναι χρήσιμη κατά με. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έννοια κατά μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζήτηση. Ε, για να καταλήξει κανεί όμω θα πρέπει να αλλάξει τη συνθήκη. Αλλά όπως λένε ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλέας, σε αυτή την κατάσταση είμαστε σήμερα. Τώρα, στα πλαίσια συνδιαλλαγής κάναμε το καθήκον μας και τηρήσαμε τις υποσχέσει μας. Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε, δημιουργήσουμε... δεν είπαμε ότι μια οδηγία ε, η οποία θα αφορά το θέμα που αφορά τη συνδυασμό επαγγελματικής και εικονιακής ζωής. Συζητάμε και αν μπορέσουμε να καταλήξουμε θα μπορούμε να, να πούμε ότι έχουμε πετύχει μια πρόοδο. Και τώρα ένα άλλο θέμα. Για το θέμα της υιοθεσία. Δεν ξέρω αν είναι θέμα γλωσσικό, δεν κατάλαβα καλά. Τι εννοείται, υιοθέτηση παιδιών, Ε, τι εννοείται για υιοθέτηση παιδιών ή ότι δέχεται κανείς κάποια πράγματα. Με ποιο... Για ποιο τρόπο χρησιμοποίησατε τη λέξη ε, έγκριση, adoption λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά ή όχι. Μήπως κάνω κάποιο λάθος, είναι μήπως γλωσσικής φύσεως. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα πλαίσιο σαφέστατα όσον αφορά το θέμα ε, ο πρόεδρος αναφέρεται στη λέξη adoption με την ιδιότητα υιοθετώ τώρα και λέει ότι ο, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι σαφέστατη όσον αφορά αυτό το θέμα. χρησιμοποίησε τη λέξη adoption που σημαίνει και υιοθεσία και έγκριση και δεν κατάλαβε ο κύριος Επίτροπος αν πρόκειται περί υιοθεσίας ή περί έγκρισης. actually, there must have been some uh, kind of misunderstanding. Εγώ δεν μίλησα για την υιοθεσία, μίλησα για την έγκριση του gender budgeting. Στην προσπάθειά μας να έχουμε πολιτικές που θα υποστηρίζουν την ισότητα ανδρών και γυναικών πρότεινα να εγκρίνουμε τη φιλοσοφία του gender budgeting και να τα χρησιμοποιήσουμε και στις εθνικές κυβερνήσεις και να τα χρησιμοποιήσουν και οι ασκούντες πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθεί πραγματικά ο τρόπος να βρεθούν τα χρήματα για να υποστηρίξουμε τις πολιτικές ισότητας δεν μίλησα λοιπόν για υιοθεσία, adoption υπό την έννοια τη έγκριση. Euh, Ευχαριστώ πολύ γιατί δεν είχα καταλάβει εγώ το, τη λέξη adoption, νόμισα ότι μπορεί να εννοούσατε και υιοθεσία. Το θέμα λοιπόν του gender budgeting Ξέρετε και η κυρία Γκριμπάουσκα ε, το συζήτησε μαζί σας και ανέλαβε δεσμεύσεις ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένα από αυτά τα θέματα. Κατά τη γνώμη μου το θέμα του gender budgeting μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό θέμα, ιδιαίτερα για, την, για το επόμενο για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Άρα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να το συζητήσουμε διεξοδικά για να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνει κάποια αλλαγή στο προσεχές μέλλον. Για το 2013 δεν είναι μακριά. Eh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη εδώ στην Επιτροπή μας και όλη την ενημέρωση που είχαμε και ευχαριστούμε για τις ε, ε, απαντήσεις που δώσατε σε όλα τα ερωτήματα, ερωτήματα που κάνανε οι σας. Εκ μέρους της Επιτροπής λοιπόν σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σήμερα εδώ και καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας και ελπίζουμε από εδώ από το κοινοβούλια να έχουμε μια συνέχεια στη συνεργασία μας αυτή με την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάλι και τώρα σταματάμε μέχρι, μέχρι τις 3 που έχουμε συνάντηση συντονιστών και η Επιτροπή μας συνεδριάζει ξανά στις 4. Ευχαριστώ για το πρωινό αυτό και θα τα πούμε το απόγευμα πάλι. Ευχαριστώ.